Uh, λοιπόν, αγαπητικοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζουμε την Επίτροπο κυρία Μπούλτ για να μας ενημερώσει για τα συμπεράσματα της ε, Γενικής Συνέλευσης του ΑΙΚΑΟ στις 7 Οκτωβρίου στο Μόριαλ στον Καναδά. Να μας ε, εξηγήσει τι αποφάσεις επήρε ε, και πώς εκτιμά τη συζήτηση της διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία. Θέλουμε να ακούσουμε τι βήματα προτίθεστε να ακολουθήσετε μετά τις αποφάσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για το μέλλον της νομοθεσίας λεγόμενης Stop the Clock που σταμάτησε τον χρόνο ε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 ισχύει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοθέσμα για το Κοινοβούλιο. Το, το περασμένο μήνα στείλαμε τρεις αντιπροσωπείες στη συνεδρία ΑΙΚΑΟ συγκεκριμένα και στη Γενική Συνέλευση για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα σας δώσουμε το λόγο για την εισαγωγή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, ε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω να σας μιλήσω μετά τη συνέλευση του ε, Μανγκάρα, όπω γνωρίζετε την περασμένη εβδομάδα ε, επιτεύθηκε συμφωνία ορόσημο για να μετριαστούν οι εκπομπές της αεροπορίας ε, στη Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ στην, στο Μόντρα. Η διαπραγματευτική ομάδα μας ε, μας έκανε περήφανος, είχα την ε, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να προείσταμε και πραγματικά πρωταγωνίστησε σε αυτή την ιστορική συμφωνία. Ε, και πραγματικά αισθάνθηκα στο πλευρό μου και παραστάτες όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους γείτονες της Ευρώπης. 191 είναι οι χώρες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και επετέφθη ακριβώς επειδή ήμασταν ενωμένοι και επειδή δείξαμε πάρα πολύ ισχυρή αλληλεγγύη. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ε, οικοδομούμε με τα θεμέλια αυτά. Επί πάρα πολύ καιρό οι εκπομπές της ε, αεροπορίας ήταν ε, κάτι το οποίο το είχαμε βάλει στην άκρη. Ε, είναι παγκόσμια μέτρα που βασίζονται τώρα στην παγκόσμια αγορά και σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, δεν πρόκειται κανείς να αλλάξει τακτική, να ανακρούσει πριν και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντονίσει την παγκόσμια δράση και είναι μια πρωτοφανή συμφωνία που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ε, διεθνή αεροπορία. Είναι η πρώτη παγκόσμια συμφωνία για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε ένα ειδικό τομέα παγκοσμίω. Θα ήθελα να τονίσω μερικά πράγματα σε αυτό το σημείο ανταποκρινόμαστε στις πολιτικές προτεραιότητες και την υπόσχεση του κυρίου Γιούνκερ, του Προέδρου μας, ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή, οικοδομούμε στα θεμέλια της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων για να ξεφύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα στις μεταφορές και δίνουμε μια στρατηγική στις εναέριες μεταφορές για μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Είναι φιλόδοξη λοιπόν αυτή η ε, συμφωνία για την αντιμετώπιση των ε, ρομεταφορών και των ε, εκπομπών τους. Ε, να σας πω και μερικές λεπτομέρειες. Τα μέτρα αυτά για τα παγκόσμια είναι πολύ ε, σημαντικά, ακριβώς επειδή είναι παγκόσμια και λαμβάνονται υπόψη οι πτήσεις ε, μεταξύ όλων των κρατών του ΙΚΑ, όπως είπαμε είναι 191 χώρες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση ε, αφορά όλες τις αεροπορικές εταιρείες ε, με τον ίδιο τρόπο. Είναι δίκαιη η συμφωνία, λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ε, στην ανάπτυξη και την οικονομική κατάσταση των χωρών και βασίζεται στην δραστηριότητα την αεροπορική και όχι στη γεωγραφία. Χώρες που δεν επηρεάζουν πολύ τις διεθνείς αερομεταφορές εξαιρούνται, όπως είναι χώρες τύπου Αφγανιστάν κλπ. Για ε, να γίνουν όλα αυτά. Ε, υπάρχουν σαφή κριτήρια που θα είναι δεσμευτικά από το 2027 και μετά. Και χαίρομαι ε, που έχουμε καταλήξει μια δεσμευτική συμφωνία. Στην πρώτη φάση, 2021 με 2026, 65 χώρες που θα συμμετέχουν εθελοντικά. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αυτών και μεταξύ άλλων 18 από τις 20 χώρες που έχουν ε, τις μεγαλύτερες αεροπορικές δραστηριότητες. Στη δεύτερη φάση, δηλαδή μετά το 2027, ε, ε, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, εκτός από τις χώρες που σας ανέφερα που έχουν μικρή συμμετοχή και σχεδόν αμεληταία. Τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και εκείνες που έχουν πραγματικά ένα πολύ περιορισμένο τομέα αερομεταφορών. Από το 2027 και μετά όλες οι μεγάλες χώρες ε, της αεροπορίας θα συμπεριληφθούν και έτσι δεν θα έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα επιτευχθεί η συμμεταχείριση όλων των ε, εταιριών. Οπότε είναι δίκαιο να αναμένουμε ότι περίπου 80% των εκπομπών ε, θα μειωθούν μέχρι το 2035, με έτος αναφοράς το 2020. Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει μια ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης και με μεγάλη χαρά την υπερασπιστήκαμε εμείς, έτσι ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνονται τα μέτρα αυτά τα παγκόσμια, να γίνονται πιο ισχυρά και ακόμα πιο φιλόδοξα. Ε, σε ευθεία σύνδεση με τη Συμφωνία του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει υποστήριξη και οικονομική και τεχνική για να ενισχυθούν οι δυνατότητες των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών, έτσι ώστε να μην μείνει καμία χώρα στην άκρη όλες οι χώρες θα έχουν υποχρέωση παρακολούθησης και αναφοράς από το 2019 και μετά. Μας βοήθησε πάρα πολύ η Συμφωνία του Παρισιού και σας ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι και εσείς παίξατε εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Επειδή η Συμφωνία του Παρισιού είναι η πρώτη πραγματικά παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα και παρά τις ε, διεθνείς ε, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρονται ρητά στη Συμφωνία του Παρισιού ούτε οι διεθνείς μεταφορές ούτε η διεθνής ναυτιλία. Και εγώ θέλω να ενταχθούν. Πάντως, ε, ο ΆΕΜΟ και ο ICAO έχουν στόχο και έχουν αναλάβει το καθήκον να το αντιμετωπίσουν. Εν πάση περιπτώσει δημιουργήθηκε τώρα ευκαιρία και με το Παρίσι για να καταλήξει ο κάο Μόντρα. Ελπίζω αντίστοιχα να ισχύσουν και για την αυτιλία. Θα είναι ενθαρρυκτικό και για άλλους κλάδους εκτός μεταφορών να προχωρήσουν σε πιο δεσμευτικές ρυθμίσεις. Η συμφωνία της περασμένης πέμπτης είναι το πρώτο βήμα για το περιορισμό της αύξησης των εκπομπών των καυσαερίων από τα αεροπλάνα θα αυξηθούν οι στόχοι, θα αναθεωρούνται και θα συμπληρωθούν από πιο μακροπρόθεσμους στόχους, πάντα σε συμφωνία με το, τα όσα αποφασίστηκαν στο Παρίσι. Όλα αυτά τα μέτρα ε, δεν πρόκειται να καλυφθούν μόνο από την παρούσα συμφωνία. Χρειάζονται και άλλα. Μεταξύ αυτών, βελτίωση της τεχνολογίας αεροσκαφών. θα πρέπει να βάλουν στόχους για πράσινες τεχνολογίες και να επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και την ε, καινοτομία. Τώρα είναι η ώρα. Δεύτερο, λειτουργικές βελτιώσεις. Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε επενδύσει ε, πολλά χρήματα στο ΣΕΖΑ, ε, στην αεροπορία είναι ένα καλό σύστημα διαχείρισης της εναέρειας κυκλοφορίας. Και Εναλλακτικέ πηγές ενέργειας για την αεροπορία τουλάχιστον στην πρώτη φάση τα βιοκαύσιμα μπορούν να παίξουν ε, σημαντικό ρόλο. Και θα ξέρετε ότι πριν από λίγες εβδομάδες η Ευρώπη λάνσαρε ε, το πρώτο παγκοσμίω αεροσκάφος που κινείται με υδρογόνο και ελπίζω αυτή η τεχνολογία να επεκταθεί. this deal in the context of the EU ε, Στα πλαίσια όλων αυτών, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2017 θα αποφασίσει για το τι μέλη γενέστε. Και τώρα εκτιμούμε, αξιολογούμε σε βάθος όλα τα ενδεχόμενα και τις δυνατότητες ε, στα πλαίσια του ETS, του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Στόχος μας είναι ακριβώς να καλύψουμε τους κλιματικούς στόχους, αλλά αυτό που μπορώ ήδη να σας πω είναι ότι υπάρχουν ήδη σαφείς αρχές για ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης, αναθεώρησης, χωρίς επικαλύψεις ε, και ένα πιο ισχυρό σύστημα στο μέλλον. Παρόλο που οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές και τελικά η επίτευξη συμφωνίας είναι επιτυχής, ε, η συμφωνία αυτή είναι ένα πρώτο βήμα και μόνο. Τώρα στο μέλλον θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα τεχνικά ζητήματα και τα εφαρμοστικά. Όλα τα τεχνικά δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα. Υπάρχει ένα πλαίσιο για τη συνέχεια, για την παρακολούθηση, για την αναφορά, για την επαλήθευση κτλ. Όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εγκαίρως για να αρχίσει να λειτουργεί η συμφωνία από το 2021 και μετά οι κανόνες που συμφωνήθηκαν στον ΑΕΚΑΟ θα πρέπει τώρα να υιοθετηθούν ε, στο ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και να εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί διεθνώς, έτσι ώστε τα όσα συμφωνήθηκαν να γίνουν πραγματικότητα. Και εδώ προσβλέπω στη δική σας υποστήριξη, έτσι ώστε από κοινού να διαμορφώσουμε τα επιπλέον βήματα για να προχωρήσουμε με τρόπο πάρα πολύ επικοδομητικό προς την κοινή ε, ατζέντα, ε, το προ... προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Οι αερομεταφορές κυριαρχούν εδώ, είναι ένας ε, τομέας που ανθεί και διατηρεί την οικονομία μας ανταγωνιστική. Έχουμε μια στρατηγική Λασάρ τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι ένα ευρύτατο σχέδιο για να αναπτυχθεί στις επόμενες δεκαετίες η ε, αεροπορία στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μειωθούν οι πτήσεις στην Ευρώπη, ούτε να είναι τόσο ακριβές ώστε να ξαναγίνουν ένα προνόμιο για τους πλουσίους. Έχουν παρέλθει αυτές οι μέρες στην αεροπορία, αλλά η συμφωνία που επετεύθη θα φέρει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτήση. Και όλοι οι ενεχόμενοι θα βρίσκονται στην ίδια μοίρα γιατί είναι παγκόσμια συμφωνία. Αξιότιμα μέλη, είμαι βέβαιη ότι ορισμένοι από εσά θα θέλατε μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών. Πιστέψτε με, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε περισσότερα και διαπραγματευόμαστε για περισσότερες και πιο φιλόδοξες λύσεις από την περασμένη φορά. Εν πάση περιπτώσει δεν ε, ξεπεράσαμε καμία κόκκινη γραμμή μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη συμφωνία αυτή με τις τεχνικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνίστησε σε αυτά τα τολμηρά βήματα, σε μια παγκόσμια συμφωνία, έτσι ώστε να αρχίσει η πολιτική αεροπορία να παίρνει αποστάσει από το διοξείδιο του άνθρακα. Ε, Σα ευχαριστώ την Επιτροπή σας και την Επιτροπή Μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω του Ευρωβουλευτές Τζούλι ε, Γκέρλινγκ και Μπα Έκχαουτ, Ελπίζω να το είπα σωστά από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον κύριο Νίλσεν, Γιάννης Νίλσεν και ε, τον κύριο Άντορ Ντέλη από την Επιτροπή Μεταφορών ε, για την παρουσία τους ε, στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μοντρέαλ. Αλλά και πολλοί άλλοι βουλευτές συνεισέφεραν από την Επιτροπή Μεταφορών και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και πραγματικά με μεγάλη προσήλωση και με πολύ στένος βοήθησαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. προς το συμφέρον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειλικρινά σα ευχαριστώ. Και το ξέρω ότι η σκληρή δουλειά είναι μπροστά μας, αλλά προσβλέπω ε, στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων και στα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε και εκεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για την εισαγωγική σας ε, δήλωση. Και τώρα έχουμε τον πρώτο γύρο παραμβάσεων με τους συντονιστές και μετά το δεύτερο γύρο τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτα, Πίτερ Λίζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Τζοβάνι. Ευχαριστώ και την Επίτροπο και όλους εκείνους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αγωνίστηκαν τόσο στο Μόντρεαλ. το πρόβλημα είναι σημαντικό. Την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο κύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού και είπε ο πρόεδρο της ομάδας μας Μάνφρετ Βέμπερ ότι αυτό θα αποτελέσει ίσω τη μεγαλύτερη πρόκληση τη ανθρωπότητα η καταπολέμηση τη κλιματικής αλλαγή. Στη συζήτηση ακούμε συχνά ότι οι αερομεταφορέ συμμετέχουν μόνο σε ένα κλάσμα των εκπομπών αλλά ε, τα πάντα είναι θέμα προοπτικής. Αν δεν κάνουμε τίποτα θα αυξηθούν οι εκπομπές. 129 χώρες, 129 χώρες είναι στη Συμφωνία Παρισιού και αν ε, αφριστούν οι εκπομπές τους, είναι όλες μαζί ε, όσο ε, οι κυκλοφορίες. Ε, Ουγγαρία, Φιλανδία, Σουηδία και μεγάλες χώρες αεροπορίας όπως το, το Κατάρ και η Σιγκαπούρη. Δηλαδή θα μπορούσε να βγει το Κατάρ και η Σιγκαπούρη και να σου πει και σιγά τι εκπέμπουμε. Εμεί δεν θα συμμετέχουμε στη συμφωνία. Όχι. Ε, δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Ο στόχο ήταν φιλόδοξο και σημαντικό πάντα για όλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μπορεί να ήταν τυχαίο, αλλά την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλη είχαμε το ψήφισμα για το Μαρακές, για την επόμενη διάσκεψη για το κλίμα και εκεί το Κοινοβούλιο αποφάνθηκε για τη συμφωνία ε, στο Μόντρεαλ και την υιοθέτησε. Ε, είναι απογοητευμένοι όλοι οι βουλευτέ, όχι μερικοί από εμά. Είπατε some of you ε, στα αγγλικά, είμαστε απογοητευμένοι. Ε, είναι απογοητευμένο όλο το κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για μείωση, δεν μιλάμε για μείωση των εκπομπών που θα χρειαζόταν για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα για του μηχανισμού αντισταθμιση έτσι, offset, αν λειτουργούν και βοηθούν το περιβάλλον και για την υπόλοιπη βιομηχανία τα έχουμε ήδη καταργήσει τα καταργούμε στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Και σε αντίθεση με τα όσα κάναμε το 2013 και ακούσαμε από τον ΙΚΑΟ, ε, όλα αυτά θα είναι δεσμευτικά μόνο από το 2027 και βλέπουμε. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, Θεέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας τα απορρίψουμε και να συνεχίσουμε στην μερίσια διάταξη και να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά ίσως και το, το πλήρες πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας, όχι. Ε, δεν θα το συνιστούσα. Μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι, θα πρέπει να οικοδομήσουμε από αυτού που έχουμε τώρα. Αρκετά δύσκολο ήταν να επιτευχθεί. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν ευκαιρίε να διατηρηθεί το σύστημα ETS στην Ευρώπη και αν χρειαστεί να μετεξελιχθεί έτσι ώστε να αποτελέσει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στη ρύθμιση αυτή stop the clock που έχουν παγώσει τα πάντα και το αρχικό πεδίο εφαρμογή. Και θα ήταν σημαντικό, κυρία Επίτροπε, να μα το επιβεβαίωσετε και πάλι. Την προπερασμένη εβδομάδα είχαμε συζήτηση μαζί σα που είπατε ότι δεν πρόκειται να ενδώσουμε εκεί σε καμία περίπτωση. Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν υπάρχει κανένα deal ε, να απεμπολίσουμε το σύστημα εμπορία εκπομπών μα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ασχοληθεί με το ETS ε, και σε ένα έγγραφο θέσεων που έχουμε μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, ε, Βιομηχανίας φέρνουμε το στόχο για τις ενδευρωπαϊκές πτήσεις να το προσεγγίσουμε στον στόχο των άλλων ε, κλάδων. Η χαλιβουργία, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερο στόχο και ο σιδηρόδρομος. Είναι στο ETS. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα της αεροπορίας. Αλλά αν μιλάμε για ποσά της τάξης των 3 σεντ, στη Χαλιβουργία και στο Σιδηρόδρομο είναι τελείως διαφορετική τάξη μεγέθους. Να το κοιτάξουμε λοιπόν και να βρούμε ε, ένα αντιστάθμισμα δίκαιο. Μπορεί να μην γίνεται αυτό αμέσως, αλλά προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αερομεταφορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο το σύστημα ITS. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να περάσουμε στο πλήρες πεδίο εφαρμογής, θα πρέπει σταδιακά του χρόνου να βρούμε μια συμφωνία για να αλλάξει η νομοθεσία. Γιατί η νομοθεσία λέει από το 2017 και πρόστιμα το 2018 ισχύει το ETS και για διπυρωτικές πτήσεις. Τώρα κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σκόπιμο, ούτε φρόνιμο, γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εθελοντικά συμμετέχουν από το 2021 και πάρα πολλοί άλλοι. Και για την Κίνα θέλω να ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, συμμετέχουν μεν, αλλά όχι απολύτως. Πού συμμετέχουν και πού δεν συμμετέχουν οι Κινέζοι. Έχω και μια ρητορική ερώτηση, δεν περιμένω απάντηση, ούτε θέλω να σας φέρω σε αμηχανία. Αλλά ας υποθέσουμε ότι Κίνα, Σιγκαπούρ, Κατάρ, Ηνωμένε Πολιτείε, αεροπορομάνες, εν περιπτώσει, με πολλές εταιρείες, από το 2021 συμμετέχουν και θέλουμε και το καλωσορίζουμε. Και μετά υπάρχουν ορισμένοι σχετικά εύποροι ως χώρες που είναι στο παράρτημα 1 στο Κιώτο και στο Παρίσι και δεν συμμετέχουν. Ποιο λόγο θα είχαμε εμείς να, πώς να το πω τώρα, έχουμε συμφωνία με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά για το ΙΚΑΟ Και με ποιο δικαίωμα θα πάμε σε τρίτες χώρες ε, όπως είναι η Ρωσία και να τους δίνουμε ένα συγχωροχάρτη και να μην δεσμεύονται να κάνουν τίποτα. Γιατί να μην μπουν στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λογική απάντηση και δεν περιμένω, αλλά να σκεφτούμε τι θα γίνει μέσω ΑΙΚΑΟ και αν, αν δεν περάσουν όλα αυτά από εκεί υπάρχει και άλλη λύση. Ευχαριστώ. η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι εδώ και που μας ανέφερε ε, τα πεπραγμένα της. Όλοι συμφωνούμε το 2016 ήταν μια σπουδαία ημέρα με τη Συμφωνία των Παρισίων και την επικαιρωσή αλλά και με τη Συμφωνία ΙΚΑΟ που ανοίγει το δρόμο για μια αλλαγή μακριά πια από, τις, από την οικονομία με εκπομπές άνθρακα. Ε, το μήνυμα είναι καλό, με κάποια κενά. Βεβαίως, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί στην αισιοδοξία μας ό,τι αφορά τη συμφωνία στην διάσκεψη ΙΚΑΟ στο Μοντρεάλ, διότι το να γίνεται αυτό ε, θελοντικά η μείωση των εκπομπών, εντάξει, έχουμε αμφιβολίες παρότι την ιστορική συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν αρκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας. Και βέβαια θα πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για να περιορίσουμε τις εκπομπές. Διότι τελικά το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές ΙΚΑΟ θα ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία των Παρισίων και βεβαίω υπάρχει και ο σκοπός, ε, ο στόχος να μειωθεί η κατανάλωση άνθρακα στο σύστημα μεταφορών. Ε, δεν πρόκειται να πετύχουμε τον στόχο για ουδετερότητα σε επίπεδο άνθρακα που προλέπεται το Παρίσι έτσι. Θέλουμε λοιπόν αυτό να είναι μια αρχή, η αρχή μιας διαδικασίας που ελπίζουμε ε, θα μπορέσει ε, να συμπεριλάβει ισότιμα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βεβαίως συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό σας, καλωσορίζουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Έχουμε ακόμα δρόμο, ε, υπάρχουν οι δικτύες ασφαλείας που αναφέρονται στο EU ETS, ε, η ΚΑΟ πρέπει να εφαρμόσει ε, κριτήρια στεναρά, εάν θέλουμε πραγματικά να περιορίσουμε στους 1,5 βαθμούς Κελσίου την θέρμανση του πλανήτη. Αναφερθήκατε επίση στα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε διεύρυνση τη χρήση βιοκαυσίμων στον τομέα τη αεροπορία να βασίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητα. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόν στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, με την αποψήλωση των δασών και των γέων ε, μόνο και μόνο για να παράγουμε βιοκαύσιμα. Ε, υπάρχουν και άλλες ζητήματα που χρήζουν διευκρίνηση. Πώς θα καλύψουμε το κενό ε, μεταξύ των φιλοδοξιών ΙΚΑΟ και των στόχων 2020-2030 του Παρισιού. Επίσης, πώς ε, τα επιζήμια ε, σε πλεονεκτήματα για τον οποιοδήποτε κλάδο. Τώρα εδώ μιλάμε για την αεροπορία. Αλλά πώς αυτά τα πλεονεκτήματα, τα επιζήμια θα μπορέσουν να παληθούν να θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε το EU ETS. Επίσης, εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι η συμπέληψη της διεθνούς αεροπορίας είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και το, σύμφωνο για το κλίμα και τις επιπτώσεις του. Θα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμα αντίσταση ε, σε μέτρα που βασίζονται στην αγορά. Εδώ προτείνεται μια φόρμουλα τεχνολογικής και επιχειρησιακής βελτίωσης, καθώς και την ευρύτερη χρήση βιοκαυσίμων για τη μείωση των εκπομπών. Ωραία, εντάξει, είναι ένα θετικό βήμα, αλλά αμφισβητούμε κατά πόσο αυτό είναι αρκετό. Καλό είναι να ξέρουμε την άποψή σας, αλλά και την άποψη της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η Julie Gerling. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπούλτς ε, και να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο της. Πήγα στο Μοντρεάλ μετά από αυτήν και άκουσα το όνομά της πολλές φορές ε, για το την προσωπική προσπάθεια που κατέβαλε. Επίσης να, ευχα... να αναφέρω την ομάδα του Χέντριν Κόλολάι, δεν ξέρω αν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Α, εδώ είναι κάποια, από την ομάδα του εδώ, εν πάση περιπτώσει. Ε, ακόμα φαντάζομαι προσπαθούν να συνέλθουν έτσι, ήταν έντονη η προσπάθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτήν το αυτό το συντονισμό, σε συντονισμένη προσπάθεια. Ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς τα κράτη-μέλη ε, ε συνεργάστηκαν ε, συντονισμένα, συνεργάστηκαν καλά, τρία χρόνια μετά τα γεγονότα που μας ε, τραυμάτισαν όλους, ε, νομίζω πως καλό είναι που μπήκε τέλος σε αυτό. Βεβαίως ε, δεν πετύχαμε ακριβώς αυτά που θέλαμε. Εμείς, όταν λέω εμείς εννοώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το ξέραμε βέβαια πριν πάμε εκεί, διότι αυτά που υπήρχαν επιτάπητο στη διαπραγμάτευση, οι κόκκινες γραμμές, δεν ήταν οι κόκκινες γραμμές που είχαμε, είχαμε θέσει πριν από 6 μήνες, ήταν ρεαλιστικές κόκκινες γραμμές μετά τη συνεδρίαση τη ομάδα φίλων τη Προεδρία και τη συμφωνία που προέκυψε από εκεί για τη διαπραγμάτευση. Και δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν δεδομένο, ε, έγιναν προσπάθειε να αλλάξουν κάποια πράγματα, ε, έγιναν προσπάθειε ε, να διαταράξουν την ισορροπία που είχαμε επιτύχει και καταφέραμε όμω εμεί να αποφύγουμε αυτέ τι προσπάθειε να τι αποκρούσουμε. Τώρα τι μα έχει απογοητεύσει. Οι δύο φάσει. το γεγονό ότι είναι μια θελοντική φάση που δεν ξεκινάει πριν από την δεκαετία του 20, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει υποχρεωτική φάση πριν από το 2027. Αναρωτιέται κανείς ε, δηλαδή τι θα γίνει. Ο ρεαλιστική, ρεαλιστικός μηχανισμός εφαρμογής ουσιαστικά θα αρχίσει να ισχύει από το 2027 και, και μετά. Οπότε αργεί ακόμα. Ε, πολλές λεπτομέρειες ε, δεν έχουν συμφωνηθεί, όλα τα MRV, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, συμφωνώ με αυτά που είπατε προηγουμένως εγώ ανησυχώ και την προσωπή μας ανησυχεί σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαφάνειας, διότι αυτή η διαδικασία για να φτάσουμε και να συνδιαμορφώσουμε αυτή την νομοθεσία θα είναι δύσκολο και σύμφωνα με τους κανόνες ΙΚΑΟ ιδιαίτερα με το καθιστό παρατηρητή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα στοιχεία που υπάρχουν κατά της δημοσιοποίησης ιδιαίτερα το ε, γεγονό ότι κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν, δεν επιτρέπεται να μοιραστούν τα έγγραφα εργασία ε, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε, ούτε μεταξύ του δεν μπορούν να μοιραστούν τα έγγραφα. Ο καθένα δηλαδή μόνο του. Αυτό ισχύει και του ΜΚΙΟ είναι μια οργάνωση έτσι αρκετά σκοτεινή, αν θέλετε, σε ζητήματα διαφάνεια. Το έχω πει και στον πρόεδρο του ΕΚΑΟ αυτό ε, και με ακούει, με, πάντα ακούει ευγενικά, αλλά καλό θα ήταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι, ποια είναι η πρόοδος που σημειώνεται σε σχέση με τα benchmarks τα οποία έχουμε θέσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα με κάποια από τα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια ήταν κάτι επί το οποίο είχαμε συμφωνήσει όλοι πριν από έξι μήνες ήταν ένα σημαντικό στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καταφέραμε. Επίσης, δεν είναι απλά μια αναθεώρηση, έτσι. Ε, είναι μια προσπάθεια προσαρμογής και βελτίωσης. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια ρητή αναφορά σε περιφερειακά συστήματα. Βεβαίω αυτό που δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία ορισμένε φορέ είναι, πιο είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που περιλαμβάνεται. Οπότε καλό είναι που έμεινε εκτό. Ε, έγινε αναφορά στην ποιότητα των offsets. Είπαμε ότι δεν πρέπει να επανεφεύρουμε τον κύκλο. Ξέρουμε πολλά ε, για την ποιότητα των offset. Καλό θα είναι η πραγματογνωμοσύνη της Ένωσης εδώ ε, να έρθει να συνεισφέρει. Θα ε, ανυπομονώ να δω το, την αξιολόγηση αντικτύπου για το σύστημα UETS. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό μαζί με την έκθεση του Ιανουαρίου ή θα μπορέσουμε να το δούμε πριν, να τη δούμε πριν την μελέτη αντικτύπου, διότι Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί βέβαια, αλλά ε, έχουμε την εντύπωση ότι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη ε, του BMGM θα είναι μικρότεροι σε σχέση με το σύστημα το οποίο έχουμε εμείς τώρα. Οπότε θα πρέπει να τα δούμε αυτά εξαιρετικά προσεκτικά. Προσωπικά νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνολική συμφωνία ε, ε, όταν κάποιος βρίσκεται εκεί ξέρετε είναι σαν παθαίνει κάποιο σύνδρομο της Στοκχόλμης έτσι ε, δηλαδή παθαίνει μια αιμονή με το θέμα αυτό ε, και μετά από κάποιες μέρες ε, όταν κοιτάζει πίσω του εμένα μου έχει μείνει μια εικονοποίηση που φτάσουμε στη συμφωνία διότι μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στο μέλλον αυτή η συμφωνία ξέρω ότι εσείς θα συνεχίσετε την προσπάθεια αλλά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση τώρα να επαναπαυθούμε είναι μόνο η αρχή έτσι λοιπόν θα συνεργαστούμε μαζί σας και με την Γενική Διεύθυνση Κλίμα που θα δώσει συνέχεια ε, στην έκθεσή μας. Αυτή η συμφωνία μας δίνει ένα πεδίο αυτή τη στιγμή ε, πάνω στο οποίο θα, κοιμηθούμε, θα κινηθούμε όπως είπε και ο Πίτερ υπάρχουν πολλές εναλλακτικές ναι, ναι, ξέρω, έχω μακρηγορήσει, αλλά τελειώνοντα να πω ότι σα ευχαριστώ πολύ για την εισφορά σα. Ξέρω ότι μπορούμε να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα ακόμα. Ευχαριστώ. Sorry, but we have... Λυπάμαι, uh, λέει ο πρόεδρο. Συμπάθημα, αλλά έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο. Κύριε Γκερμπράντι, πρώτο. Ευχαριστώ, πρόεδρε και κύριε επίτροπε που ήρθατε. Και σας ευχαριστούμε για το έργο που έχετε επιτελέσει. Βέβαια, τα υπόλοιπα που θα ακούσετε θα είναι επικριτικά. Όμως πιστεύω ότι χωρίς ε, τα όσα κάνατε, χωρίς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είχαμε κλείσει αυτή την συμφωνία. Θα πρέπει για τη σύναψη αυτή να είμαι θα υπερήφανη. Και ξέρετε, δεν ξέρω αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Πάντως γεμάτο δεν είναι σίγουρα. Οπότε, οπότε συζητούμε για την ε, κλιματική αλλαγή. Πολλές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα και οδυνηρά. Οπότε τότε χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Δηλαδή τι ισχύει για την αλλαγή του κλίματος πραγματικά. Να, να σας πω έτσι κάποια στοιχεία Εάν θέλουμε να μείνουμε κάτω από το 1,5 τότε έχουμε περίπου 5 χρόνια μπροστά μας. Αν πάμε στο 2 στους 2 βαθμούς έχουμε μεταξύ 10 και 30 χρόνια μπροστά μας. Αυτά με τις ε, σημερινές εκπομπές. Άρα ασκούμε πίεση σε όλη τη βιομηχανία για να περιορίσει τις εκπομπές. Στον αφορά τώρα ε, την αεροπλοεία, και περιορίζουμε την αύξηση. Όχι μόνο την ε, περιορίζουμε, αλλά και έχουμε και το συμψηφισμό, την αντιστάθμιση, που δεν είναι περιορισμός, δεν είναι μείωση. Τι αποσπάσαμε στο Μοντρέλ. Η ΚΑΟ είχε δεσμευτεί το 2013. Δεν τηρήθηκε η υπόσχεση εκείνη. Με τίποτα δεν υπάρχει ε, αύξηση διοξιδίου του άνθρακος ουδέτερη. Άρα ούτε καν αυτό που υποσχεθήκανα δεν τηρούν οι δυσικά. Και αντίθετα ήταν πάρα πολύ κοινικό το ότι μετά τα πανηγύρια για το κλείσιμο της Συμφωνίας των Παρισίων δεν ήμασταν σε θέση να κλείσουμε μια συμφωνία που να πλησιάζει, το να συμβαδίζει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι στην Ένωση, συγκεκριμένα στο Κοινοβούλιο, είμαστε πολύ στριμωγμένοι. Πώς θα αξιολογήσουμε αυτή τη συμφωνία, τι θα κάνουμε με, τις, το σύστημά μας, το, το σύστημα των εκπομπών και της εμπορίας του, στο ETS. Καλά, έχουμε και άλλα στοιχεία τώρα. Η ποιότητα του offset, του συμψηφισμού, τέλος πάντων. Πάντως, έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η ισχύ ότι στην φάση τη προαιρετική μπορεί ακόμη να αυτοεξαιρεθούν μέσα σε αυτήν την εξαετία κάποιες χώρε. Δηλαδή, αν περάσει ένα χρόνο, μετά να αποφασίζουν ότι δεν του αρέσει η συμφωνία, μπορούν να βγουν, να μπουν ξανά κλπ. κλπ. Δηλαδή κάποιο εκούσια προσχωρεί και δεσμεύεται μετά ή ου. Επίσης όσον αφορά την ε, Κίνα. Αυτό που σημαίνει και δεν είναι και τόσο στεγανό. Δηλαδή δεν ευθυγραμμίζονται 100% με αυτό το οποίο εμεί ορίζουμε ω ανάπτυξη, ω αύξηση. Νομίζω είναι σημαντικά αυτά τα δύο σημεία, αν μπορείτε να τα σχολιάσετε. Ευχαριστώ κύριε Σέικαουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και εσάς κύριε Επίτροπε που ήρθατε και για το ότι σωστά προφέρατε το όνομά μου. Πολύ σπουδαίο αυτό. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, γιατί νομίζω ότι εδώ έχει δημορφωθεί κάποια συνένεση. Συμφωνούμε στο πώς αξιολογείται η συμφωνία αυτή και από πλευρά ΣΥΚΑΟ και από πλευρά κλίματος. Ε, πρόκειται για δύο πράγματα που απήχαν έτη φωτό το 2013 κουβέντια η Ευρωπαϊκή για αλλαγή του κλίματο, αλλά νομίζω ότι στι συναντήσει με το ΙΚΑΟ δεν λέγανε ούτε κουβέντα. Ήταν ε, κάτι το οδυνηρό αυτό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μάθημα επόδυνα. Οπότε είδατε τρόπος πήγε το πράγμα στην κουβέντα του 2016. Η αλλαγή του κλίματος ήταν παρούσα, ήταν, ήταν βασικό θεματολόγιο και, από παντού, από, τα νησιά του Μάρσαλ, από την Μπουρκίνα, Φάσο, Γουατεμάλα, έξω από τα δόντια το είπαν. Όλοι αυτοί γιατί, γιατί νιώθουν την αλλαγή. Άρα δεν είναι πια ακαδημαϊκή κουβέντα. Για αυτές τις χώρες είναι κάτι πολύ χειροπιαστό. Οπότε αυτό ήταν πολύ διάκριτο. Και έτσι άλλαξε όλη η κουβέντα με την ΙΚΑΟ. Και Καλά τα λέει η Τζούλια όταν μα τα λέει στη μητρική τη γλώσσα που μα είπε ότι είναι ένα οργανισμό που δεν έχει καμία διαφάνεια, μα είπε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι παλιωμοδίτικος οργανισμό. Έτσι θα τα λέγει ένα Ολλανδό που μιλάει Αγγλικά. Τέλο πάντων, πριν από κάνα χρόνο ούτε κανεί θα τολμούσε να βάλει πόδι, να πατήσει μέσα στο δωμάτιο αν ήταν ε, οικολόγος, αν ήταν πράσινο, Ενώ ξέρουμε ότι αυτές οι επαφές, αυτές οι συζητήσεις είναι εξεχόντως πολιτικές. Ο ΙΚΑΟ έχει προϊστορία, αλλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν πολλά. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια αν θέλουμε να έχει αξιοπιστία στο μέλλον η κάθε επαφή. Θα έχουμε πολλά θέματα που ακόμα πρέπει να συζητηθούν. Ε, άρα για όλα αυτά πρέπει να γίνουν με διαφάνεια. Πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω όμως ότι ακόμα το έχουν χωνέψει ή του ΙΚΑΟ. Να και λένε κιόλα από τη Συνεκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή πριν την Ολομέλεια, αυτοί που ετοιμάζουν την Ολομέλεια λοιπόν, άλλωστε η Ολομέλεια μεταδίδεται στο ίντερνετ, η Εκτελεστική λοιπόν Επιτροπή και εγκλεισμένων των θυρών τα λέγανε και, και παραπονιόντουσαν γιατί κάποιοι ε, χρησιμοποιούσαν tweet. Μα ήταν διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος να ξέρει κάθε χώρα τι πρεσβεύει. Τι πρεσβεύει. Δεν ήθελαν οι να υπάρχουν tweets να μην ξέρουν τι γίνεται, τι, τι, τι λένε, τι προσβεύουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλει ο ΙΚΑΟ να αποκτήσει αξιοπιστία και να τους εμπιστευόμαστε, χρειάζεται να ασπαστούν την διαφάνεια. Τα είπαν λοιπόν οι περισσότερες και σας τα ρωτήσανε σωστά. Ε, όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε εκείνο το ψήφισμα για το ε, MBM, τη συμφωνία, τι που ισχύει, αλλά έχουμε και σε ένα άλλο ψήφισμα ε, το τι θέση έχουμε για, τη, για, το, για τους στόχους των εκπομπών. Και η Ρωσία και η Ινδία επιφυλέχθηκαν για το παγκόσμιο MBM, την Παγκόσμια Συμφωνία, αλλά και η Κίνα και η Αργεντινή και η Βενεζουέλα, αλλά καλά εντάξει. Τι σημαίνει επομένω αυτό, σημαίνει ότι η Κίνα ακόμη δεν έχει χωνέψει τι θα ισχύσει μετά το 2020 δεν έχουν ασπαστεί, δεν, ε, δεν έχουν χωνέψει ότι πρέπει να δεσμεύονται για αυτόν τον στόχο. Τι θα γίνει επομένως μακρόπνο με το στόχο. Καλά έχουμε την ε, ε, τριετή αξιολόγηση και αναθεώρηση, αλλά αυτό είναι πιο πέρα, πιο μακριά. Τώρα, ε, βλέπω ότι σηκώνει το σφυρί ο πρόεδρος, οπότε θα ολοκληρώσω. Αυτά για τα όσα κάναμε με τον ΙΚΑΟ. Πρέπει να κάνουμε και άλλα εδώ, στην Ευρώπη. Αυτά πήγαινε στο Μόντρελ ήταν απλώς ένα θεμέλιο, μια αφετηρία. Πάνω σε αυτήν θα πρέπει να συνεχίσουμε, να χτίσουμε. Παντού βλέπουμε ότι για την ε, αεροπλοεία γίνονται πολλά. Στον Καναδά γίνεται κουβέντα για το διεξίδιο του άνθρακα. Ε, συζητάνε και για τις αεροπορικές μεταφορές. Συζητάνε για εκπομπές στην Κίνα και εκεί ασχολούνται με την αεροπλοή και τις μεταφορές, άρα τα πράγματα αλλάζουν. Ε, καιρός ήταν. Άρα καιρός είναι και η Ευρώπη να κάνει κάποια βήματα. Τα είπαμε για το ETS, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και για τη δράση που θα λάβουμε στο μέλλον, έτσι, σε αυτή την ε, εσωτερική αγορά όπως τη λέμε. Άρα καλά, εντάξει το Μόντρεαλ, αλλά να δούμε και εδώ και τα του οίκου μας. Είπαμε μπήκε το θεμέλιο και να μην χτίσουμε πάνω στο θεμέλιο όπως θα ήθελε ε, η βιομηχανία. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Οι συντονιστές μίλησαν ε, πεντάλεπτο, επτάλεπτο ο καθής. Οπότε τώρα έχουμε λιγότερο χρόνο για τους συναδέλφους. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε με τις ε, ερωτήσεις και κατόπιν με τη να απαντήσει η κυρία Μπούλτσα. Ήβο, Ήβο Μπέλετ, σε παρακαλώ, περιορίζω στο δίλεπτο ή δυνατόν. Θα προσπαθήσω. Γεια σας, Επίτροπε, καλώς ορίσατε. Είχε το Bloomberg ένα ρεπορτάζ την περσμένη εβδομάδα και έλεγε για μια πτήση Καζαμπλάνκα Μαδρίτη. Το κόστος το 2030 θα ήταν 50 δολάρια έως 130 για την πτήση αυτή. Έτσι λέει το Bloomberg. Άρα 31 cents έως 80 cents ανά επιβάτη. Ε, δεν είναι και τόσο φιλόδοξη συμφωνία επομένως. Πάντως αυτό συμφώνησε ο ΙΚΑΟ, τα είπε ο κύριος Λίζε και θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες και της βιομηχανίας για να μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο του 40% λιγότερες εκπομπές με στόχο του 2030. Αλλά όχι μόνο οι άλλες βιομηχανίες αλλά και η αεροπλοεία θα πρέπει να το φροντίσει αυτό. Τι εγγύσεις υπάρχουν. Είναι ο μηχανισμός των offset στεγανός. Πώς είστε σίγουροι ότι τα δικά μας πρότυπα θα τα ασπαστούν. Το Μάιο με επικεφαλή στην Τζούλη πήγαμε και εμείς τα είπαμε εκεί πέρα. Ακριβώς η έλλειψη διαφάνειας μας εντυπωσίασε. Εγκρυπτό και απαραβίστο δουλεύουν θα έπρεπε να έχουν περισσότερη διαφάνεια. Πλήρη διαφάνεια. Ε, αυτό και θα τους ε, ζητήσουμε. Να σεβαστούν την αρχή της διαφάνειας στο μέλλον. Παρακαλώ, εσείς διαβιβάστε το μήνυμα αυτό στον ΙΚΑΟ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Νίλσον. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήμουν και εγώ παρόν στο Μοντρεάλ εκπροσωπώντας την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οφείλω να πω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και το Συμβούλιο, όχι μόνο Κομισιόν και Κοινοβούλιο, πολύ καλή συνεργασία είχαμε. Και αυτό ήταν καλό σημάδι. Ότι μπορούν να συνεργάζονται τόσο αγαστά Καλά, εμείς βασικά ήμασταν παρατηρητές. Τα κράτη-μέλη ε, έχουν το βασικό λόγο ε, και στον ΙΚΑΟ, αλλά αξίζει να ποτίσουμε φόρο τιμής στα κράτη-μέλη. Γιατί κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μιλήσει με μία φωνή. Έκανε πολύ καλή δουλειά το Συμβούλιο. Αλλά και εδώ τελικά επετύχαμε αυτή την ιστορική συμφωνία την οποία και καλωσορίσαμε. Είναι όντως ιστορική. Για πρώτη φορά έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για τέτοια θέματα. Όπως σας είπα όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Αλλά όπως είπανε και άλλοι συνάδελφοι και άλλα κράτη, τα επόμενα χρόνια θα πρέπει αυτό το σύστημα να το οικοδομήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μακροπρόθεσμα, βιώσιμο και αξιόπιστο γιατί τελικά τι θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και ε, για καινοτομία, βιοκαύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Για να το καταφέρουμε αυτό, και αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι σπουδαία συμφωνία. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Ωραία. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις όμως που θα πρέπει να απαντήσουμε και να συζητήσουμε. Μια που έχετε έρθει στην Επιτροπή μας, κύριε Επίτροπε. Η στρατηγική για την αεροπορία, ο κανονισμός για την ΕΑΣΑ, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ, κυρία Φώστερ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είναι εδώ η Επίτροπος, αλλά και η ομάδα, η Είδαμε και τον κύριο Χόλαντ χθε στην Επιτροπή Μεταφορών να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και τρία χρόνια. Κάποιοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, μεταξύ των οποίων ο Πίτερ Λίτε, ο εισηγητή, τουλάχιστον δέκα χρόνια. Έτσι λοιπόν για πολλού εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά θέλουμε απελπισμένα να βρεθεί ε, μία λύση, να φτάσουμε σε μια κατάληξη για αυτό το θέμα. Τώρα κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά το αρχικό σύστημα που ήθελε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το, παλιό EUTS δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί. Ήταν, δημιουργούσε πολλές αντιπαραθέσεις, ήταν πολύ περιοριστικό, θα δημιουργούσε τεράστιες τρευλώσεις ανταγωνισμού και δεν υπήρχε επαρκή πολιτική βούληση ε, για να μπορέσει να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής Τρεν, Τραν πήγε την προσωπή μας στο Μοντρεάλ και στην Οτάβα το Μάιο ο συνδυασμός αυτών των επισκέψεων βοήθησαν. Αυτό που σωστά αναγνωρίζει ο επίτροπο είναι το θέμα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δηλαδή που θα βοηθήσει να λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι έχουν ε, εμπειρία από την αεροναυπηγική, την, ε, το διάστημα, την ε, τεχνολογία του διαστήματος και γίνεται προσπάθεια εδώ και καιρό να προχωρήσουν σχέδια όπως το Clean Sky 1-2, ε, το Cesar ε, και η υποστήριξη που υπάρχει από τα θεσμικά όργανα πρέπει να συστηθεί επ' αυτού. Η ανησυχία, μου, η ανησυχία μου είναι ότι εντάξει, ωραία, ε, το ΙΚΑΟ δεν είναι τέλειο, κανένα θεσμό, κανένα θεσμικό όργανο δεν είναι τέλειο, ο καθένα έχει του κανόνε του, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να πούμε ε, ε, πώς θα αλλάξει η δομή της ΙΚΑΟ. Δεν, προ, δεν, δεν θα αλλάξουμε την δομή της ΙΚΑΟ. Το βασικό είναι να έχουμε μια καλή σχέση συνεργασίας με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, για να μπορέσουν να προχωρήσει τη διαδικασία. Ε, τα υπόλοιπα είναι χάσιμο χρόνο. Επίσης ανησυχώ κάπως, ε, και δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, αλλά ένας συνάδελφος αναφέρθηκε σε μια συμβαστική λύση, να φτάσουμε σε ένα συμβασμό λίγο από το παλιό EU ETS ε και λίγο, από το μέλλον. Όχι, θα ήταν τεράστιο λάθος αυτό εάν τα μέλη αυτής της Επιτροπής, η Επιτροπής Τραν, θεωρούν ότι μπορούμε τώρα ε, να γυρίζουμε πίσω το χρόνο και να πάμε πίσω στο σύστημα που είχε προταθεί αρχικά, διότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είτε θα ακολουθήσουμε αυτήν την οδό, ε, και δεν το λέω συχνά κυρία Πίτρο, πραγματικά πιστεύω ότι έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Εμείς συχνά επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πραγματικά ε, κάνατε τεράστια δουλειά και εσείς και τα κράτη-μέλη υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία και η άποψή μου είναι ότι εάν δεν συνεχίσουμε σε αυτό, σε αυτό το δρόμο είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτός ο δρόμος πολύ μεγάλη ευκαιρία για να λύσουμε το θέμα των εκπομπών. Και αυτό το κοινοβούλιο θα μπορούσε αυτό να το καταστρέψει. Σε αυτή την επιτροπή, σε μια άλλη επιτροπή, θα μπορούσαμε πραγματικά να το τορπιλήσουμε. Να μην το κάνουμε, παρακαλώ. Διότι αν δεν φτάσουμε σε συμφωνία αυτή τη φορά, δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε σε συμφωνία. Και χαίρομαι που όλοι συμμετέχουν στη διαδικασία, που παίζουν το παιχνίδι. Παρότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των μεγάλων χωρών, αλλά κάποια στιγμή ε, θα ακολουθήσουν, διότι είναι προ συμφέρον του. Σα ευχαριστώ λοιπόν για το έργο σα και σίγουρα θα έχετε τη συνεργασία, ελπίζω, όλων των μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις επιτροπές. Εγώ θα κάνω σίγουρα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να δώσω μια όθηση σε αυτό το εγχείρημα και να σας υποστηρίξω όσο χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην σας κάνω να χρησιμοποιήσετε το σφυράκι. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Ξέρουμε ότι έκανε σκληρέ προσπάθειε, πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει. Ευχαριστούμε και όλου του συναδέλφου που είχαν πάει εκεί και τον προσπάθησαν. Πραγματικά είναι ιστορικά αυτά, ε, το είπαν και άλλοι. Στην COP21 κανεί δεν περίμενε να ε, υπογράψουν όλοι. Καλά, εντάξει. Η υπογραφή δεν σημαίνει και έργα και για τον ΙΚΑΟ είπα ότι εντάξει κάτι θα βγει, αλλά είχα τι επιφυλάξει μου αν αυτό που βγήκε θα λειτουργήσει. Τώρα, Φυσικά δεν είναι αυτό που θέλαμε εμείς, σε καμία περίπτωση είναι σαφές αυτό. Χαίρομαι για τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί φοβόμουν ότι θα φάμε πολύ ξύλο, ε, επειδή δεν τα θέλαμε έτσι, θα τα κάνουμε μόνοι μας και διαφορετικά. Πάντως αυτό το αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι προαιρετικό και εθελούσιο, ε, αξίζει την υποστήριξή μας. Και θα μπορούσα να φανταστώ, εφόσον υπάρχει κάθε τριετία ρήτρα αναθεώρησης, είναι και φιλόδοξο. Γιατί ε, για τον 1,5 βαθμό, για το COP21 το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αν σκεφτώ και την πολιτική για τους ωκεανούς και τις θάλασσες που ασχολούμαι πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να καταστραφούν τα κοράλια αν αυξηθεί η θερμοκρασία του νερού κατά 1,5 βαθμό. Ε, και να κάνω και ερώτηση τώρα. Είπαμε ότι υπάρχει υδρογονοκίνητο αεροσκάφος πλέον και γίνεται και έρευνα να χρησιμοποιούνται και άλλα καύσιμα στο μέλλον. Επίσης, ε, να υπάρχουν αεροπλάνα που στο έδαφος ε, όταν τροχοδρομούν να είναι ηλεκτροκίνητα για να κάνουμε οικονομία. Ε, και στην ναύση πλοία ε, υπάρχουν και τερματικά για τη χρησιμοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ε, και πολλά κρατημέλη τα έχουν ήδη όλα αυτά ρυθμίσει και εφαρμόσει. Πώς ε, σκέφτεστε να αλλάξουμε νοοτροπία και να ασκούμε διαφορετικά και πολιτική. Υπάρχει δυνατότητα και έδαφο εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίμωβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και σα κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ να μα παρουσιάσετε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε. Νομίζω ότι ακούσατε ε, έτσι αυτά τα λόγια εκτίμησης για το έργο σας. Τα αξίζετε. Θέλω όμως ε, να ε, φανώ και λίγο επικριτικός. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό δεν αρκεί, ότι χρειαζόμαστε να πάμε παραπέρα. Ποιο είναι το σχέδιο για να έχουμε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας και τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει για να συνεισφέρει τα επόμενα χρόνια στη διαμόρφωση των λεπτομεριών της συμφωνίας προς ωφελός μας. Επίσης, είμαι κάπως επικριτικός ό,τι αφορά το σχέδιο του να συνεχίσουμε την όθηση της ανταγωνιστικότητας ε, της ε, βιομηχανίας μας ε, της αεροναυπηγικής, διότι αν κάποιος μπορεί να μη σεβαστεί τη συμφωνία κάθε θελοντική περίοδο, αλλά και τη μη θελοντική περίοδο, τότε αυτό θα είναι δύσκολο ως πρωταγωνιστικότητα για τον κλάδο μας. Τι σκοπεύετε να κάνετε, θα συνεχίσετε να σπρώχνετε, να πιέζετε ε, και πώς αυτό θα μεταφραστεί στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Εγώ προέρχομαι από τη Σουηδία ε, και δεν είναι το ίδιο να είναι κάποιος ε, βουλευτής να έχετε από τη Σουηδία και να έχετε το Λουξεμβούργο. Έρχομαι 13 ώρες με το τρένο, δεν γίνεται να έρθω από τη Σουηδία, καταλαβαίνετε. Πώς λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτό στην εσωτερική αγορά, πώς θα συνεχίσουμε με μια καλύτερη συμφωνία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αν θέλω να μου πείτε τι είδους ε, σχέδια ε, έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Κάλεμπαχ είναι τελευταία, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια παράκληση έχω από όλη αυτή τη συζήτηση, διότι σε παρελθόν ε, τα έχουμε ξαναδεί. Σας κατανοώ και σας προσωπικά για τη διαπραγμάτευση και όλους τους παρόντες ότι ήταν τεράστια επιτυχία και βγαίνετε και προς τα έξω και το πανηγυρίζετε Ε, και καλό είναι αυτό και υγιές για τον άνθρωπο έτσι να ε, τα κάνει όλα αυτά. τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά μπορεί να είναι και ένα ηρεμιστικό και ένα καταπραϊντικό φάρμακο. Θέλει προσοχή αυτό. Μην τρελαθούμε από τη χαρά μας τώρα και ε, δεν προσέξουμε. Είναι ένα πρώτο βήμα. Μην ξεχάσουμε να δουλέψουμε να ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε βάλει με τη Συμφωνία του Παρισιού. Δηλαδή, για μας έχει σημασία να πούμε σήμερα ότι μπράβο μας, πετύχαμε κάτι σπουδαίο, αλλά παραμένουν τόσα πολλά ανοιχτά θέματα που θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά και να σταματήσουν οι πανηγυρισμοί. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα να λάβει το λόγο η Επίτροπος Μπούλτς για να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις. Για να ξεκαθαριστούν οι απορίες που υπάρχουν για τη συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενθαρρυντικά όσα είπατε. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προόδου και είμαι βέβαιη ότι δεν θα με αφήσετε να ξεκουράζομαι στις δάφνες μου. δεν ήταν πάντοτε βέβαια αποθετικά όσα είπατε, αλλά νομίζω ότι όλα όσα άκουσα θα με βοηθήσουν. Άρα ε, θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή, νιώθουμε την πίεση που μας ε, ασκείται, αλλά νομίζω ότι ο διάλογος ε, πρέπει να είναι επικοδομητικός, δηλαδή να τα συζητούμε και να βρίσκουμε λύσεις. Ακριβώς για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας επίσης και για να ε, συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά ε, αυτόν τον ε, τομέα και όχι μόνο στην αεροπορική βιομηχανία αλλά και στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Οπότε ακριβώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την απασχόληση που έτσι ανεβαίνει και λοιπά και Τέλος πάντων να σας απαντήσω σε ό,τι μπορώ και αν κάποιος θεωρήσει ότι δεν καλύφθηκε, σε έρθει σε επαφή μαζί μας ε, και θα το απαντήσουμε γιατί θα πρέπει αμέσως να φύγω τώρα γιατί έχουμε κάλλη ε, υποχρέωση μια άλλη συνεδρίαση για τη χρηματοδότηση των ε, μεταφορών πρώτα πρώτα για το ETS η πρώτη δέσμη ερωτήσεων ακόμη εξετάζουμε όλες τις επιλογές τίποτα ακόμα δεν έχει κλείσει και να σας πω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες σήμερα κάνουμε αυτή την πρώτη συζήτηση σε κάποιο άλλο θεσμικό όργανο, κατόπιν έχουμε συνάντηση στο Συμβούλιο. Και θα πάω τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο για αυτό το λόγο. Θα συναντήσω την κυρία Κανιέτη εκεί τη συνάδελφο και έχουμε τώρα για τη συμφωνία, για το MBM, τη συμφωνία. Θα δούμε τι θα γίνει από το 2017 Βέβαια και θα γίνει και αξιολόγηση επιπτώσεων. Αυτό θα γίνει επίσης από τον Ιανουάριο του 2017 και θα συζητηθούν όλες οι επιλογές. Σίγουρα έχουμε κατά νου πάντα τις βασικές μας ε, αρχές, τους στόχους σχετικά με το κλίμα. Ε, αυτά τα οποία πάγια θα συζητούσαμε. Οπότε για αυτές τις κόκκινες γραμμές τις οποίες ε, σεβαστήκαμε, τις στηρίσαμε και ε, έτσι θα συνεχίσουμε. Είστε επικριτικοί για το ποιος συμμετέσχε. Όπως είπατε για την Γουατεμάλα, ήρθαν και άλλα μικρά κράτη. Μα ακριβώ γι' αυτό ήρθανε. Γιατί θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία. έτσι αποκτούν σπουδιότητα. Άρα υπάρχουν πολλά κίνητρα. Αυτό θα ισχύσει για όλους όσοι δεν έχουν μπει ακόμα στο ETS. Μέχρι σήμερα έχουμε 65 χώρες που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα. Ε, βέβαια και εγώ θέλω περισσότερες. Ε, ελπίζω να έχουμε ακόμη περισσότερες. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν καν αρχίσουν διαπραγματεύσει διαβεβαίωσε τις χώρες αυτές πώς έχουν τα πράγματα και είπε ότι θα τύχουν βοηθείες που την χρειάζονται. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα γιατί εύκολο είναι να βάζει κανεί δύσκολους στόχους αλλά αν δεν έχω τα εργαλεία, τα μέσα επίτευξη αυτών των στόχων ε, τότε δεν έχει κανένα κανένα δυνατό χαρτί στα χέρια του. Αλλά εμείς όμως δείξαμε ότι έχουμε τα μέσα να πετύχουμε. Βιομηχανία, τεχνολογία, τους είπαμε. Ε, ρωτήθηκα επίσης για το τι είδους τεχνολογία. Νέα συστήματα, νέα υλικά. Νέοι τρόποι οργάνωσης. Βιοκαύσιμα. Μέχρι τότε θα έχουμε πάει στην τέταρτη γενιά. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα βάλαμε στην στρατηγική μας για την απαλλαγή από το διοξίδιο και στο πρόγραμμα της μεταφοράς. Επομένω είχαμε και τις μεγαλύτερες χώρες, είπατε και για Ρωσία και Κίνα και περιμένουμε η Κίνα πλήρως να συμμετάσχει. Θα συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα τους Κινέζους εδώ στις Βρυξέλλες. Και πάγια τους τα λέμε και συνεχώς τους προσκαλούμε. Επίσης, μόνο έξι ήταν οι χώρες που δεν προσυπέγραψαν αυτή την συμφωνία για το διοξίδιο. Άρα, τώρα όλοι μαζί πιέζουμε τις υπόλοιπες χώρες. Άρα μόνο έξι από τις 191. Τώρα, σαν αφορά ποιοτικά στοιχεία των offset, είναι σημαντικό Παραλαμβάνω ότι θα πιέσουμε για την υπόθεση αυτή τα ποιοτικά offset και τις τεχνικές συζητήσεις. Αυτό που ήδη καλύψαμε ήταν να έχουμε μια διακυβέρνηση ποιοτική. Πολύ σημαντικό. Ό,τι και να είναι οι χώρες ή οι εταιρείες, εμείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Για τη φιλοδοξία, μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη συμφωνία δεσμευτική σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας. Έχουμε το 80% των εκπομπών που αυτή τη στιγμή καλύπτονται. Άρα σας εκλυπαρώ, βοηθήστε με να βάλουμε τον πύχη ακόμη πιο ψηλά. δεν θα ξεχάσουμε το στόχο. Θα μας απασχολεί συνεχώς. Δεν φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Συνεχίζεται η διαδρομή προς την υλοποίηση. Πάμε για... μετά το 2027. για τις νέες τεχνολογίες και θα πρέπει να, παρακάμψουμε όλους τους φραγμούς για να κόψουμε το διοξίδιο που δημιουργείται από τις αεροπορικές μεταφορές. Ε, πολύ δαπανηρά όλα αυτά. Βλέπετε, εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα με, μεγάλο. Επίσης, είπατε για την διαφάνεια. Εγώ θα εξασφαλίσω ότι θα συνεχίσετε να εμπλέκεστε όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω. Πάντοτε θα έρχομαι όταν με καλείτε. Το είπαμε στην ΙΚΑΟ. Πιστεύω ότι πήραν το μήνυμα και θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Βιοκαύσιμα. Είναι σημαντικό συμμετρικά να προχωράει κάνει για όλου τους τομείς. Αλλά βέβαια εδώ πέρα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Είπαμε είμαστε σε δεύτερη, τρίτη γενιά, αλλά ελπίζουμε ότι με τα βιοκαύσιμα στην τέταρτη γενιά θα προχωρήσουμε. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι 44 όλοι προσπάθησαν για να αποσπάσουμε ό,τι γινόταν. Και στο μέλλον θα γίνει αυτό. Α, κάτι άλλο που δεν σας το είπα, αλλά πρέπει. Είπαμε με τον κύριο Κανιέτε, τα πάμε πολύ καλά, συνεργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, συντονιζόμαστε. Και αυτό ήταν ένα δυνατό χαρτί που είχαμε. Ήταν αυτή η συμμαχία με φιλόδοξους στόχους. Ε, αυτό ήταν ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο προς ε, όλο τον κόσμο. Εγγύησες, Αγαπητέ συνάδελφε, όσες θες να σου πω, όπως για όλα τα θέματα της ζωής, τόσο πολλές. Αλλά είναι φιλόδοξη η στόχη για την αλλαγή του κλίματος για αυτή την ουδέτερη αύξηση των εκπομπών. Μα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις αερομεταφορές, ισχύει για όλες τις μεταφορές. Είδατε και με την βιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια, για τα ηλεκτρικά οχήματα τέλος πάντων και προχωράμε βλέπετε ολοταχώς με την ενέργεια, με τα αεροδρόμια πλοία. Είδατε και για τα αεροδρόμια θέλουμε να υπάρχει ουδετερότητα για το διοξίδιο. Ε, νομίζω ότι οι μεταφορέ επιτέλου ανταποκρίθηκαν. Ότι θα πρέπει να ανανοιάζονται για το περιβάλλον. Φυσικά ποτέ δεν είμαστε στο 100% αλλά κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μα. Ε, κάποια στιγμή θα έρθει άλλος να με διαδεχτεί και θα κάνει ακόμα περισσότερο. Εγώ πάντως θα έχω εξαντλήσει τις δυνατότητες μου. Και συμπερασματικά σας επαναλαμβάνω. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει η συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Να χρησιμοποιούμε επικοδομητικά τις επικρίσεις, την εξέβρεση λύσεων. Και συνέχεια να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Εγώ ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα πολλά και αύριο περισσότερα και θα πρέπει να συνεχίσετε η προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Άρα το θέμα θα μείνει ζωντανό, το συζητάμε και εσείς συνεχίστε να μας πιέζετε, να μας προκαλείτε. Εμείς θα αντιδράσουμε. Το ETS μας προσδίδει κάποια αξιοπιστία. Είναι μοχλός για να πετύχουμε πολλά στη διεθνή φόρα. Θα καταφέρουμε πολλά σε παγκόσμιο κλίμα, το ξέρουν όλοι. Μας παίρνουν στα σοβαρά και για αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν έξω από το παιχνίδι καμία χώρα να μην μείνει απ' έξω. Θα αρχίσουμε και τις επενδύσεις. 44 δις πρότεινε για τις γειτονιάζους χώρες της Αφρικής. Και έτσι να έρθουν και αυτοί να μπουν στις διαπραγματεύσεις. Και αυτοί στο θέμα των μεταφόρων. Άρα λιθαράκι, λιθαράκι, σε όλα τα επίπεδα θα καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή να πετύχουμε αυτού του φιλόδοξους στόχους για την αλλαγή του κλίματος, το κλιματικό θεματολόγιο. Μαζί, μαζί θα προχωρήσουμε. Χέρι-χέρι θα τα καταφέρουμε. Σα ευχαριστώ και για τις επικρίσεις και τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε εμείς κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και σα ευχαριστώ για τι εξηγήσει που μα δώσατε για μια σειρά αποζητήματα. Σα ευχαριστούμε που απαντήσατε στα ερωτήματα των συναδέλφων. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην εμείς διάταξη. I invite Mr. Corbett. Και τώρα ο κύριος Κόρμπετ να προσέλθει παρακαλώ για να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο. First Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόρμπετ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας έτσι ώστε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μας για τη γνωμοδότησή μας που ψηφίζουμε. Σας παρακαλούμε να μας παρουσιάσετε τις σύντομες αλλά τις βασικές μάλλον αλλαγές που προτείνεται ε, για την τροποποίηση του κανονισμού μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα των διοργανικών ε, διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών σε δεύτερη ανάγνωση. Ε, Δήμερο συζητήσαμε διάφορα θέματα σήμερα το πρωί και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω κάτι που έχει να κάνει με την τροπολογία 265 που φαίνεται μάλλον προβληματική για τη δεύτερη ανάγνωση. Οι διαπραγματεύσεις δεν βασίζονται πια στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στην κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Άρα, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, που τροποποιεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα καλύψει θέματα ε, που συμπεριλαμβάνονται στη θέση του Συμβουλίου, ούτε θα μπορεί να αντιδράσει ε, ε, όσα προσεγγίζει το Συμβούλιο. Επιτρέπει λοιπόν το άρθρο 69 να αποκλίνουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μας λοιπόν αυτό να γράφεται και ε, στο άρθρο 73 εδάφιο γ του κανονισμού. Και η απόφαση μιας επιτροπής να αρχίσει διαπραγματεύσει, θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία έτσι ώστε να είναι διαφανής η διαδικασία. Και αυτά που λέει η τροπολογία 265 ε, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε τεχνική ε, νομοθεσία με τέτοιο τρόπο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κόρμπετ, πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι μετά τη διμερή συνάντηση που είχαμε σήμερα, αναδιατυπώσαμε κάπως τη συμβαστική τροπολογία έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και η άποψη του κύριου Κόρμπετ και τα σχόλια του και τη στείλαμε στους συντονιστές. Αρχές του απογεύματος, νωρίς το απόγευμα. Συγγνώμη, αλλά ο χρόνος πίεζε πάρα πολύ. Δίνω μέσα το λόγο στον κύριο Κόρμπετ για να μας εξηγήσει τη θέση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε είναι χαρά μου που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι αυτή η Επιτροπή είναι ε, πραγματικά στην πρώτη γραμμή ε, μια σειρά θεμάτων όταν είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ε, το Ευρωκοινοβούλιο απέκτησε το δικαίωμα στην απόφαση, τότε λοιπόν η ομάδα περιβάλλοντος και η ομάδα προστασίας καταναλωτών ε, αυτές οι επιτροπές ήταν που ε, προώθησαν τις διάφορες τεχνικές για να εκμεταλλευτούμε τη διαδικασία ε, συναπόφασης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των θεσμών. Έχετε, έχετε δηλαδή μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά τις σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η έκθεση μου για τη γενική αναθεώρηση του οικονομισμού καλύπτει μια σειρά από είναι ε, αποτέλεσμα δύο ετών, εργασία δύο ετών, όπου σε, μια ομάδα που συμμετείχαν όλες οι πολιτικές ομάδες, ε, ε, υποστήριξε και μια task force όπου οι, γραμματείε όλων των επιτροπών εκπροσωπήθηκαν. Είναι λοιπόν κάπω διαφορετική αυτή η έκθεση από τι άλλε, όπου απλά ο εισηγητή παρουσιάζει ένα κείμενο, όλοι οι υπόλοιποι που βάλουν τροπολογίες και μετά διαπραγματευόμαστε μια συμβαστική λύση. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση μου είναι το αποτέλεσμα δύο ετών συμβιβασμού κατά την ε, προετοιμασία αυτού του κειμένου. Ελπίζουμε λοιπόν να περάσει χωρίς πολλές αλλαγές, αλλά εκεί βεβαίως που θα χρειαστεί ε, θα ακούσουμε προφανώς. Ένα σημείο κλειδί στο οποίο αναφερθήκατε. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων πριν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, μετά την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο, μετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έχουμε εντύπωση λοιπόν όταν γίνονται διαπραγματεύσει. Είναι προφανέ ότι το σημείο αφετηρία για αυτέ τι διαπραγματεύσει είναι η θέση του κάθε θεσμικού οργάνου κατά την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο αφετηρία. Όλοι γνωρίζουμε ότι στι διαπραγματεύσει πρέπει να βρεθεί ένα συμβιβασμό. Το λέει και η συνθήκη. Το λένε οι κανόνες μας. Τριμερής διάλογος, διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Και όλοι πρέπει να μετακινηθούν από την αρχική τους θέση. Καλό θα ήταν βεβαίω να μετακινούνταν μόνο το Συμβούλιο, αλλά ε, δεν συμβαίνει αυτό συνήθω. Όταν λοιπόν λέμε ότι η εντολή είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, δεν αναμένουμε οι διαπραγματευτέ να πούν αυτή είναι η θέση μας, ε, δεν θα μετακινηθούμε». Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, πάντα μετακινούμαστε από τη θέση μας. Αλλά το σημείο αφετηρίας είναι αυτό που ε, ψήφισε η Ολομέλεια. Δεν μπορούμε στους κανόνες μας να πούμε ότι οι επιτροπές μπορούν να επιλέξουν ένα διαφορετικό σημείο αφετηρίας και να αγνοήσουν αυτά που έχει εγκρίνει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε ε, είναι να λέμε ότι όταν η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει νέα στοιχεία που δεν καλύπτονται από τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, τότε η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγματευτική ομάδα. Δηλαδή η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τη κάποια νέα στοιχεία και να δώσει κάποιες οδηγίες σε επίπεδο επιτροπή, χωρί να χρειάζεται να ξαναπάει δηλαδή στην Ολομέλεια τα, τώρα τι, τι όταν λέμε νέα στοιχεία, δεν είναι κάποια προσθήκη στο κείμενο ε, διατύπωσης, είναι ένα νέος παράγοντας, ένα νέο στοιχείο πολιτικό, πραγματικά καινούριο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να δώσει νέε οδηγίε στη διαπραγματευτική ομάδα, ούτως ή άλλως ε, τα μέλη της ίδιας της Επιτροπής είναι αυτά που διαπραγματεύονται. Ε, οπότε είναι στενή η αλλω τα μελη τη ίδια τη επιτροπης ειναι αυτα που διαπραγματευονται οποτε ειναι στενη η σχεση και από εκεί πέρα θα ακολουθείτε στην σημερινή διαδικασία, ε, τριμερή διάλογο, οι διαπραγματευτέ του Κοινοβουλίου επανέρχονται, δίνουν αναφορά στην Επιτροπή, λένε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε θέση εδώ, αλλιώ θα φτάσουμε σε συμφωνία. Εκεί όμω πρέπει να αντισταθούμε στεναρά, δεν πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο θα υποχωρήσει και στο τρίτο θέμα ε, θα φτάσουμε στον τάδε συμβιβασμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρόθεση ε, στο κείμενο αυτό. Μετά τη συνάντηση που είχα νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρό σα, τον κύριο Λαβία, σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ο κανόνας αυτός, να βελτιωθεί το κείμενο, εν πάση για να καταστεί σαφέστερο. Να μην αναφερόμαστε μόνο στη θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, αλλά να λέμε ότι αυτό υπόκειται και στον κανόνα 69, στον οποίο μόλις αναφερθήκατε, που καθορίζει τα κριτήρια για να μπορέσει κάποιο να απομακρυνθεί από την θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Εάν αν έγιναν εκλογέ παραδείγματο χάρη μετά την πρώτη ανάγνωση. Να λάβουμε υπόψη μα το αποτέλεσμα ε, των εκλογών, έτσι, φυσιολογικό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό θα το διευκρινίσουμε λοιπόν στο κείμενο, υπάρχουν και κάποια άλλα, κάποιες άλλες ε, τροποποιήσεις διατύπωσης, αλλά νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί επαρκέ και θα γίνει αποδεκτό ε, το κείμενο αυτό από την Επιτροπή σας, αλλά και από άλλες Επιτροπές βέβαια. Αυτά ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Πρέπει να πω και το έχω πει και νωρίτερα ότι μετά τη συνάντηση σήμερα το πρωί μετά τα κατάσταση γραμμές οδηγίες λέμε ε, συμπεριλαμβανομένων και υπό τη υπό τη μορφή τροπολογιών, τροποποίησεων. Ναι, συγγνώμη να επαναλάβω, δεν ήταν το δικό μου μικρόφωνο αναμένο. Ε, μετά τη σημερινή συνάντηση, λέω, έχουμε προσθέσει άλλο ένα σημείο. Μετά τον όρο guidelines, τι γραμμέ ακόμα και υπό τη μορφή τροπολογιών έχουμε προσθέσει για να γίνει σαφέστερο πώς θέλουμε να εργαστούμε για να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής της ομάδας διαπραγμάτευσης ε, που είναι, και μέλη της Επιτροπής. Επάσε ανοίγει τώρα η συζήτηση. Ε, ο κύριος Τόρβαλτς έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ρίτσαρντ που ήρθε εδώ. Στην Επιτροπή αλληλία. Ε, βρήκαμε τρόπους, βρήκαμε μάλλον και ένα κοινό τόπο και νομίζω το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσαμε να βρεθούμε εδώ στην Επιτροπή Ένβη. Είπατε πολύ ωραία προηγουμένως ότι η Επιτροπή Ένβη είναι κατά κάποιο τρόπο ο προπομπός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. εγώ μετά τις εκλογές έλαβα το φάκελο iLook. Η υπόθεση αυτή, το θέμα αυτό, ευθύς εξ αρχής, ήταν κοινή ε, ευθύνη, κοινή ε, αρμοδιότητα ένβη και επιτροπών ένβη και Και αυτό περίπλεξε τα πράγματα. Η ήτρε στην δεύτερη ανάγνωση είχε μείνει κάπω απ' έξω. Αλλά για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να περάσει ο φάκελος ε, και μετά τον τρίλογο να φτάσουμε στην αποτέλεσμα δηλαδή υπήρχε μια διαρκή συζήτηση με αυτούς που ήταν εκτός και αν δεν, μπορούσαμε, αν δεν είχαμε μπορέσει να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις τους ε, πιθανότατα μπορεί και η δεύτερη ανάγνωση να μην είχε πάει καλά. Ξεκινάω λοιπόν εδώ στην ε, μεικτή αρμοδιότητα, κάτι που συμβαίνει συχνά εδώ. Πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολος είναι ο τριμερής διάλογος σε δεύτερη ανάγνωση. Πώς μπορεί να γίνει δύσκολος, όπως περιπτώσει. Ταυτόχρονα ήταν εξαιρετικά τεχνικό το συγκεκριμένο θέμα. Περίπλοκο. Είχαμε δύο οδηγίε εξαιρετικά τεχνικές και οι δύο, όπου ακόμα και μια αλλαγή διατύπωση μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Ήταν δύσκολο, όπω περιπτώσει. Και από ιδεολογική πλευρά ήταν δύσκολο το θέμα. Διότι διάφορες πολιτικές ομάδες, ακόμα και αν έγιναν εκλογές ε, στο ενδιάμεσο, ε, οι πολιτικές ομάδες ε, είχαν πολύ σαφή και έτσι άτεκτη άποψη για, τα, για το ζήτημα. Όταν λοιπόν δημιουργούμε κανόνες που, δυσκολεύει, που δυσκολεύουν την προσπάθεια να ληφθούν υπόψη όλα αυτά και όλες οι απόψεις, κάποιος που είναι εκτός της φούσκας αυτής, θα πει καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτό είναι, αυτός είναι ο κίνδυνος εδώ. Δεν θα ήταν βέβαια καταστροφή, αλλά θα ήταν επιζήμιο για τη δημοκρατία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις αυτές, να δημιουργήσουμε δηλαδή κανόνες που είναι τόσο περιοριστικοί, τόσο στενοί, που δεν δίνει τη δυνατότητα ε, να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Έπρεπε να δω και Φρεντερίκ Φρίς, ε, η Φρεντερίκ Φρίς για να σας πει τη δική της άποψη, γιατί και αυτή είχε αναλάβει με τέτοιο φάκελο στη δεύτερη ανάγνωση, με τέτοια υπόθεση, αλλά τρέχουμε από εδώ και από εκεί, το ξέρετε και εσείς προσωπικά, ε, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Αυτά πάντως εν συντομία, αυτή είναι η άποψή μας, οπότε η προσέγγισή σας ε, είναι εξαιρετικά σημαντική για μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η Τζούλη Γκέρλιν. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ένα άλλο σενάριο. Να σας πω, η κυρία Κάτεμπαχ ήταν η συγγήτρια τότε. Ε, επεκτάθηκε σε δύο κοινοβουλευτικές θητείες πριν και μετά τις εκλογές και είχαμε δυσκολία για την εντολή. Ήταν ένας κανονισμός πλαίσιο στη δική μας Επιτροπή που ουσιαστικά επηρέαζε τις διαπραγματεύσεις για ένα άλλο νομοθέτημα σε άλλη Επιτροπή. Ήταν εδώ ε, ο κανονισμός για τα τρόφιμα και στην Επιτροπή Γεωργίας για τη βιολογική γεωργία. Είχαμε σαφή ε, εντολή ενώ εκείνοι στην Επιτροπή Γεωργίας ε, είχαν και αυτοί δώσει εντολή και πήγαν την έκθεσή τους στην Ολομέλεια. Και συγκρουστήκαμε σφόδρα ε, για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η συγγήτριά μας κατάφερε με τρόπο πάρα πολύ ε, αριστοτεχνικό να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Αλλά υπάρχει αρχή εντολών γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι η δική μας εντολή ήταν πιο ισχυρή ε, που πήγε στην Ολομέλεια, μάλλον δική μας έκθεση πήγε στην Ολομέλεια, η άλλη έκθεση πήγε μόνο στην Επιτροπή Γεωργίας. Υπάρχει εδώ κυριαρχία εντολή. η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, θα ήθελα να ε, σας ρωτήσω κάτι. Είχα το ε, προετοιμάσει και μεγάλη τοποθέτηση, αλλά δεν θα την κάνω. Ε, Κατανοώ τις προσπάθειές σας να επιταχυνθούν οι νομοθετικές διαδικασίες στο Κοινοβούλιο. Έχω όμως την εντύπωση ότι αυτό θα εξυπηρετήσει κυρίως τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και μικρότερες που μπορεί να αντιμετωπίζουν ε, άλλα προβλήματα και να εκπροσωπούν άλλες απόψεις, δεν θα υποφεληθούν. Διάβασα δύο συμβιβαστικές προτάσεις και έχω την αίσθηση ότι η ευελιξία μιας ε, κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, περιορίζεται προς όφελος της Ολομέλειας. Ναι, αλλά και στα μέλη ε, αυτό τι επιπτώσεις έχει. Υπάρχουν κάποια μέλη που έχουν διαφορετική άποψη στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Είναι σαν να μας λέτε κάντε ό,τι θέλετε στις επιτροπές και στην Ολομέλεια θα το κανονίσουμε εμείς. Για το συμβασμό 1β, τι σημαίνει για σας λοιπόν αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Κατευθυντήριε γραμμές λέτε μια επιτροπή. Πόσο δεσμευτικέ είναι. Μπορεί να τις αλλάξει μια κοινοβουλευτική επιτροπή στη συνέχεια. Γιατί ε, από το συμβιβασμό αυτό έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε τα χέρια μας δεμένα στο μέλλον και θα μπορούσαν να λαμβάνονται κάποιες ε, μέρμηνε για κάποιες συμφωνίες με τρόπο αδιαφανή. Λοιπόν, πρώτο, τι γίνεται με την ψηφοφορία αυτή στην και στι Ολομέλειε και τι γίνεται με την κατευθυντήρια αυτή γραμμή. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κόρμπετ, θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω ότι τι κάναμε ε, σήμερα το πρωί. Ήταν σαφής αναφορά στο άρθρο 69 του κανονισμού. Χρειάζεται σαφή ε, θεώρηση για ε, να δούμε όλα τα σημεία στη διαπραγμάτευση. Επίσης, είχαμε και μια τροπολογία ακριβώς για να γίνουν σαφείς οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες και να μην υπάρχει μόνο μια πρόταση από το διαπραγματευτή από την Επιτροπή και κατά την άποψή μα αυτό είναι καλύτερο από την προηγούμενη πρόταση. Καλά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόρμπετ να μας τα εξηγήσει αυτά καλύτερα. Ποια είναι η θέση σα και η απόψη σα. Well, thank you very much. Κόρμπετ, σα ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρατε. Και πρώτα πρώτα να σας πω για τι εκθέσεις που αφορούν δύο θητείε. δηλαδή που σας τις κληροδότησε η επόμενη ε, θητεία. Έχουμε ήδη τη διάταξη υπαριθμών 69 του κανονισμού που λέει ότι σε ΑΒΓ ε, συνθήκες και προϋποθέσεις μπορεί το Κοινοβούλιο να αποστεί από την, ε, από την πρώτη συνάντηση της πρώτης ανάγνωσης. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει η πολιτική ισορροπία δημοκρατικό. Οπότε υπ' αυτούς τους όρους υπάρχει η ελευθερία του να διαφοροποιηθεί κανείς από την τοποθέτηση της πρώτης ε, ανάγνωσης. Τώρα, τι γίνεται όταν έχουμε συναρμοδιότητα με άλλη επιτροπή. Ε, αυτό σε κάθε φάση κάποιας διαδικασίας ε, γεννά πολλά ζητήματα. Είναι περίπλοκο, είναι φυσικό. Ό,τι και να κάνετε όμως για να τα βρείτε με την άλλη επιτροπή, καλώς το κάνετε αρκεί όμως να μην αντιφάσκει με την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ή στην πρώτη ανάγνωση. Σήμερα όταν τα συζητήσαμε είπαμε α, σαν παράδειγμα το εξή. Ας πούμε λέει το Κοινοβούλιο ότι κάτι θα πρέπει να πάει στο 75% και λέει το Συμβούλιο ότι πρέπει να είναι 25%. Η εντολή για τους διαπραγματευτέ είναι να ξεκινήσουν από το 75% και να συμβιβαστούν στο βαθμό που χρειάζεται για να αποσπάσουν συμφωνία. Όμως, αυτό που δεν μπορεί να το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να πει όχι, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει από το 90. Οπότε η αφετηρία είναι η θέση του Κοινοβουλίου αυτή που εγκρίθηκε. Μέχρι την ε, τιμή, μέχρι τη θέση του Συμβουλίου. Εκεί σε αυτά τα πλαίσια κινείται η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το το περιθώριο λίγο. Δεν υπάρχει επιταγή εν λευκό. Ούτε βέβαια υπάρχει περιορισμό που κανεί να είναι σκληρό, που κανεί να είναι δεκτικό κλπ. Οπότε κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να υπερβείτε την θέση της πρώτης ανάγνωσης. Ελπίζω ότι αυτό σας δίνει να καταλάβετε τι εννοώ. Φυσικά και πρέπει ο κανονισμός να διευκολύνει το έργο μας. Εννοείται. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε μία διάταξη, ένα άρθρο στον κανονισμό που να λέει ότι μία επιτροπή μπορεί να αγνοήσει τα αποφασιστέντα στην Ολομέλεια. Ε, βέβαια, εσείς δεν κάνετε τέτοια πράγματα, αλλά κάποιοι ίσως θα το ήθελαν αυτό. Να πει, ας να λένε, εμείς θα κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το Κοινοβούλιο αποφάνθηκε... Να, αυτό είναι η απάντηση στην κυρία Γκίρλινγκ. Η εντολή της Ολομελίας εννοείται ότι κάτι ισχύει από θεσμικής. Άρα, εδώ κολλάει κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με τον κανονισμό, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις της πρώτης αναγνώσης. Όταν μια επιτροπή ξεκινάει τον τριγωνικό διάλογο, τον τριμέρι διάλογο σε πρώτη ανάγνωση, αφού έχει εγκρίνει την έκθεσή τη, αλλά πριν κατέβει η έκθεση στην Ολομέλεια, τότε αυτή η απόφαση στο μέλλον θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια. Οπότε έχουμε μια περίοδο 24 ωρών για τις ενστάσεις. Εάν υπάρξει ένσταση, γίνεται ψήφο. Ναι ή ου. Να πάμε διαπραγματεύσει ή να μην πάμε. Εάν όχι, τότε γίνεται η πρώτη ανάγνωση κρίνεται στην Ολομέλεια και μετά διαπραγματεύσει. Οπότε έτσι παρέχονται οι εγγύησει ότι αν δεν υπάρχει ένσταση τότε η Επιτροπή έχει την σιωπηλή συνένεση της Ολομέλεια και αυτό την νομιμοποιεί ακόμα παραπάνω για τις διαπραγματεύσεις. Και δεν μπορεί κανεί να το αμφισβητήσει αυτό. Κύριε Κανιέτσινα. Όχι, δεν πρόκειται περί συνωμοσία υπέρ των μεγάλων. Όταν κάναμε την αναθεώρηση του κανονισμού, συμμετέσχουν οι πάντες και οι ανεξάρτητοι βουλευτές τότε. Ή μη εγγεγραμμένοι τέλος πάντων. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να ρίξουμε κανέναν. Προσπαθούμε να είναι πιο εύρυθμη η μία εγγεγραμμένη τελο παντων οχι οχι δεν θελουμε να ριξουμε κανεναν προσπαθουμε να ειναι πιο εύρεθμη η λειτουργια του Κοινοβουλίου. Και αυτό διότι εάν αποφαίνεται για κάτι το κοινοβούλιο, η φωνή του είναι πιο δυνατή από τη φωνή μιας συγκεκριμένης επιτροπής. Αλλά είπαμε τι ισχύει για τι διαπραγματεύσει. Αυτό που είπε ο πρόεδρο, πολύ σημαντικό για τη δουλειά το είπε και ο κύριο Τόρβαλτ. Πολύ σημαντικό αυτό για ε, την ε, ε, δουλειά σα στην πράξη. Οπότε όταν έχουμε τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και αποσπούμε ένα αποτέλεσμα, τότε ποιος θα κάτσει να πει «Α, μα δεν ξέρω αν ήταν σωστή διαδικασία για τις καθημερινές γραμμές για αυτό που κάνατε». Ε, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Κατευθυντήριες γραμμές είναι. Οι οποίες υπάρχουν για να σας δίνουν και ευελιξία, ακριβώς όπως είπατε. Και πολλές φορές οι καθημερινές γραμμές οδηγούν σε συγκεκριμένες τροποποίησεις. Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά λέμε τώρα για τροποποίησεις στην θέση του Συμβουλίου. Καταλάβετε, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γνέφει καταφατικά. Ελπίζω ότι είναι σαφές. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Τόρβαλτς. Ναι, ένα ερώτημα το 75-85% στο οποίο αναφερθήκατε ως παράδειγμα. Όταν εδώ μετά μιλάμε για ένα αριθμητικό στοιχείο, είναι εύκολο να πούμε, εντάξει, αυτή είναι η θέση της Ολομέλειας, αυτό το ποσοστό έχει ψηφίσει, αλλά ορισμένες φορές οι διατυπώσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες. Και το τι βρίσκεται εντός και τι βρίσκεται εκτός της εντολής δεν είναι τόσο ξεκάθαρο σε σχέση με το παράδειγμά σας. Αυτό είναι, αυτή είναι η ανησυχία μου. Όταν δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, όταν δεν έχουμε απλά αριθμητικά στοιχεία, αλλά έχουμε ασαφείς διατυπώσεις, τι κάνουμε. Συγγνώμη, δεν σας είδα προηγουμένως για το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να μιλήσω προηγουμένως, όχι, δεν είναι ότι δεν με είδατε. Αλλά θέλω να αντιδράσω σε αυτό που ακούσαμε τώρα και εγώ μη εγγεγραμμένος είμαι, δεν είμαι μέλος κάποιας αντιπροσωπείας, μιλάμε για ένα θεωρητικό τώρα θέμα. Δέχεστε ότι εμείς είμαστε τμήμα ενός αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου. Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν παίρνουμε αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρα, αλλά κάθε ευρωβουλευτής έχει κάποια ευθύνη. Και όχι μόνο έχει ευθύνη, αλλά δικαιούται κιόλας να λαμβάνει αποφάσεις συμμετέχοντας στην Ολομέλεια. Σε ένα εθνικό κοινοβούλιο, όταν συζητούμε για την υγεία, δεν έρχονται οι γιατροί να ψηφίσουν. Ή όταν συζητάμε για τον προπολογισμό, δεν ενέχονται οι οικονομολόγοι. Οι βουλευτές αποφασίζουν. Όταν μιλούμε λοιπόν για αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι κάτι που αφορά έναν και μη επαΐοντα. Και όταν μια πολιτική ομάδα παίρνει ε, ε, ένα κατάλογο ψηφοφορίας, θα πρέπει να αποφασίζει με έναν τρόπο ε, υπεύθυνο. Δεν αποφασίζουν οι ειδικοί, καμιά φορά αποφασίζουν και μη ειδικοί. Και σε κάποιες περιπτώσεις όπως είναι η Ολομέλεια, βεβαίως αυτή δίνει εντολή πολύ πιο ισχυρή από ότι μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η Επιτροπή μας ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμησή της. Και έχετε δίκιο, αν πει Μέλια 40% για κάποιο στόχο, δεν θα πρέπει εμείς να βάζουμε το 50% ως στόχο, θα πρέπει να δεχτούμε την απόφαση της Ολομέλειας. Έτσι δεν είναι, που είναι ισχυρότερο όργανο του Κοινοβουλίου από ότι εμείς. Ευχαριστώ. Thank you very much. I don't know if you... Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε και σε αυτό. Πάρα πολύ σύντομα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τόρβαλτς για το ε, παράδειγμα που ε, έδωσα με αριθμούς είναι πιο εύκολο, είναι πιο δύσκολο όταν μιλάμε για κείμενα. Αλλά από αυτό το γεγονός και μόνο φαίνεται ότι είναι δύσκολο οποιοδήποτε να ισχυριστεί ότι ε, έχουμε αποστεί από την αρχική μας θέση. Αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Άρα αυτό υπερασπίζετε τη δική σας θέση. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων για να διευκρινίσουμε κάποια θέματα ε, που έχουμε ενώπιόν μας και για τα οποία θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα μια στιγμή. Ε, θα ψηφίσουμε αύριο, είπαμε εδώ στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 7-8 Νοεμβρίου. Η ΔΕ Ολομέλεια το Δεκέμβριο, έτσι έχει προγραμματιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει εδώ αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο. Uh, το επόμενο θέμα είναι ανταλλαγή πληροφορικών για ένα σύστημα προειδοποίηση και εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με νέε ψυχοτρόπε ουσίε. Η συγκητή μα είναι ο Κρίστιαν Μπουσόη, στον οποίο και δίνω μέσω στο λόγο για να μα παρουσιάσει το θέμα του. Uh, for uh, giving Μας πει λοιπόν την άποψή του για το σχέδιο γνωμοδότησης. Λοιπόν, οι ψυχοτρόπες ουσίες, ψυχοδραστικές, ψυχοδραστικές ουσίες ε, διακυβεύουν την υγεία των ανθρώπων, οδηγούν σε θανάτους ε, εκατομμυρίων ανθρώπων ε, κάθε χρόνο. Είναι ένα σημείο ανησυχία ε, για όλους. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι υπάρχουν έτσι ψυχοτρόπες ουσίες που όταν τις παίρνει κάποιος, ε, όταν μπαίνουν στο σύστημα το ανθρώπινο, τότε επηρεάζουν όλες τις λειτουργίες του. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια σημαντική αύξηση στον αριθμό, τον τύπο και τη διαθεσιμότητα των MPS σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο σημαντικός αριθμός των 101 ουσιών που έχουν εντοπιστεί για πρώτη φορά μέσω του συστήματος έγκαιρης το 2014 είναι εντυπωσιακό. Η σημαντική αύξηση των MPS είναι ε, ένας λόγος ανησυχίας. Όχι μόνο ε, για την αντιμετώπιση και την πρόληψη, ε, αλλά και σε επίπεδο τοξικολογίας. Η πρόταση της Κομισιόν έρχεται σε μια στιγμή όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική αύξηση στον αριθμό των διαθέσιμων MPS στην αγορά των ναρκωτικών πάνω από 500 ουσίες ε, παρακολουθούνται το διπλάσιο ε, σε σχέση με τις διεθνείς συμβάσεις. Ε, η νέα πρόταση έχει ως σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμοστεί ένα σύστημα έγκαιρης προεδοποίησης, να ενισχυθεί μάλλον το σύστημα και να υπάρχουν ε, διαδικασίες που να επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική και γρήγορη δράση. Προσπάθησα να βελτιώσω το κείμενο, να διατηρώντα την ίδια κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους για την υγεία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τη έκθεση, αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια με βάση τι νέε πιχοδραστικέ ουσίε. Πολλά έχουν γίνει για να βελτιωθούν τα στοιχεία και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα παρακολούθηση των ναρκωτικών και να ξεπεράσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσει ε, υπερεθνικέ. Ε, εξακολουθεί όμως το φαινόμενο της χρήσης NPS να αυξάνεται και αυτό είναι η πραγματική πρόκληση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και μεθοδολογικές και ε, θεωρητικές ασυνέπειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που οδηγούν σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν στρατηγικές γρήγορε παρέμβαση ή σχέδια δράσης μακροπρόθεσμα. Θεωρώ ότι όταν συζητάμε πώς, το πώς θα αξιολογήσουμε τους κινδύνους για την δημόσια υγεία θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη και τι πληροφορίε που έχουν να κάνουν με την τοξικότητα του NPS και στοιχεία σχετικά με τη διάδρασή του με άλλες ουσίες και, και προϋπάρχουσες ε, ασθένειες. Δεν είχα πολύ χρόνο. Θα υποβληθούν και κάποιε νέε τροπολογίε που θα αφορούν την ασφάλεια ε, και τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και τις σχετικές αξιολογήσεις αναμένω ε, συνεργασία με του κοινού εισηγητέ, η συνάδελφη Γραμματεία και εγώ θα οργανώσουμε μια πρώτη συνεδρία στου κοινών εισηγητών το συντομότερο δυνατόν και θα επανέλθουμε με νέε πληροφορίε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I don't know who... ευχαριστούμε, λέει ο Θέλει κανεί τον λόγο. Συνάδελφε, ο κύριος Σελίμοβιτ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, Ξεκινώ λέγοντα ότι όσο και αν αυτό είναι δευτερεύον για την Επιτροπή μα, νομίζω ότι παραμένει σημαντικό γιατί όλοι όσοι έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία ε, γνωρίζουν ότι τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με το ίντερνετ και μετά σαν έφηβοι ξέρουμε πώς προχωρούν. Οπότε ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Είναι καλή αφετηρία για να προχωρήσουμε. Επίσης αυτοί οι δείκτες που υπάρχουν λένε ότι δεν υπάρχει κανένας ε, είδους επιβράδυνση στο μέτωπο των ε, ψυχοδραστικών ουσιών. Το αντίθετο τώρα πολλούνται ελεύθερα, θεωρούνται θεμητό υποκατάστατο της ε, μεθαδόνης, της κοκαίνης, της κανάβιος και βέβαια με το ίντερνετ είναι ακόμα πιο εύκολη η διακίνηση από τις τρίτες χώρες μπορούν να έρθουν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νομικό πλαίσιο είναι φτωχό και ανεπαρκές. χρησιμοποιούν τεχνικές μάρκετινγκ και πωλήσεων και έτσι παρακάντουν το ισχύον δικαίωμα. Άρα θεωρούνται φυσικά προϊόντα, ε, φυτικά, και ε, αλλού λένε ότι ο, αυτά είναι μόνο για έρευνα, δεν είναι για κατανόηση από άνθρωπο, ούτως ώστε να μπορούν να παρακάμψουν πάλι την ε, νομοθεσία. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζω ότι ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη τον Απρίλιο του 2014, κάτω από τη Επιτροπή, έκανε ένα ψήφισμα. Το Συμβούλιο όμω καμία θέση δεν έχει υιοθετήσει. Έτσι όπω είναι τα πράγματα, επομένω, πιστεύω ότι αυτή η νομοθετική πρόταση που τώρα συζητούμε πρόκειται να διορθώσει τα πράγματα όσον αφορά το σύστημα γης για αυτές τις ουσίες και τις νέες ψυχότοπες ουσίες. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλει το λιθαράκι στην Επιτροπή μας και να βοηθήσει την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που είναι συναρμόδια. Επίση, σα τονίζω τα εξή. Αυτέ οι ψυχοενεργέ ουσίε βεβαίω αφορούν πάρα πολλά προϊόντα και θεωρούνται αυτέ τι ψυχοενεργέ ουσίε ε, προϊόν που πολλούν τα καταστήματα που πουλούν βιταμίνες, άλλοι θεωρούν ότι είναι χημικέ ουσίε έρευνα. Ε, ότι είναι μέσα για επιστημονική έρευνα ή ότι είναι ναρκωτικά διασκέδασης τέλο πάντων. Και έχουν βρει διάφορε πρωτότυπε ιδέε, πρωτότυπα ε, πακέτα, συσκευασία που λύνονται από το Ιντερνετ. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανεί να αναγνωρίσει, να διακρίνει ε, όλη αυτή την, την και την ποικιλία. Επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρήσει ότι όταν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για τεκμηρίωση της βλάβης ότι πρέπει να παρέμβει. Ναι, οπότε απογορεύει κανεί ένα προϊόν και βγαίνει ένα καινούριο. Να μην είμαστε αφελεί. Εξαπλώνται πάρα πολύ γρήγορα αυτέ οι ουσίε στην αγορά. Σε μερικέ περιπτώσει υπάρχουν ε, πάρα πολύ περιορισμένα επιστημονικά συμπέρασματα για ποιο προϊόν. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει ταχαίως να ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε φορά να αποφασίζει το αν θα απογορεύσει ή όχι. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αυτό το σύστημα ε, και θα πρέπει να ανακοινωθεί στον κόσμο. Το ξέρει ο κόσμος. Θα πρέπει να το ξέρουν οι νέοι. Το 2014 είχαμε 101 προειδοποιήσεις για ουσίες που προηγουμένως δεν είχαν απασχολήσει το σύστημα. αναδύονται έτσι ξαφνικά και πάρα πολύ γρήγορα και εξαφανίζονται πάλι γρήγορα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον κόσμο όσον αφορά αυτές τις νέες ουσίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Κονέτσνα. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης, γνωμοδότηση καλύτερα, προτάσεις κάνει. Στι νέε λοιπόν ψυχοτρόπες ουσίες, οι ψυχοδραστικές, εδώ αγωνιζόμαστε, παλεύουμε με ανεμόμυλους. Είναι χαμένη η μάχη. Ή τουλάχιστον ε, ας προσπαθήσουμε να μειώσουμε ε, τον κίνδυνο από τις ουσίες αυτές, γιατί για να τις ε, ξαλείψουμε αυτό αποκλείεται. Μετά από ολόκληρες εβδομάδες έρευνας απαγορεύονται κάποιες ουσίες και διότι έχουν αποδεδειγμένα βλαβερές συνέπειες για την υγεία, αλλά στο μεταξύ ε, οι έμποροι ε, έχουν ε, αναπτύξει άλλες 50 νέες ουσίες που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Και εμείς ενόμαστε και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και πίσω από τους διακινητές των ναρκωτικών. Δεν την κερδίζουμε αυτή τη μάχη. Πάντως, δική μας ε, ευθύνη είναι και θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, είναι λέω, Ευχαριστώ τον εισηγητή. Να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να είναι πιο ευέλικτο. θα πρέπει να πάσα στιγμή να μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον είμαστε σε θέση εγκαίρως να δρούμε, να εντοπίζουμε αυτές τις ουσίες και να προειδοποιούμε τα γειτονικά μας κράτη. Καθώς έχουμε ελεύθερη αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, οι ουσίε αυτές εντάσσονται στα συγκεκριμένα, να προειδοποιούμε τα άλλα κράτη-μέλη. Αν θέλετε να σα δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, που δείχνει ε, ότι καμιά φορά κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ε, υπάρχει μια ψευδοεφεδρίνη που χρησιμοποιούν καμιά φορά ε, φαρμακευτικές εταιρείες στην ευρωπαϊκή αγορά και κυκλοφορούν νόμιμα. Από αυτές τις ουσίες στην Τσεχία φτιάχνουν περβετίνη κρίσταλ μεθ, κρυσταλλική μεθαδόνη, που το κάνουν μετά από βρασμό αυτού του προϊόντος. Τουλάχιστον αυτή η δραστική ουσία καταφέραμε στο μεταξύ ε, ε, να μην ε, πωλείται ελεύθερα στην Τσεχία και τα σχετικά φάρμακα, που υπάρχουν και τέτοια φάρμακα, γιατί παίρνουν τα χάπια, τα βράζουν κανονικά και βγάζουν κρυσταλλική μεθαδόνη, ένα θετικό ναρκωτικό. Αυτή λοιπόν η δραστική ουσία που λέγεται εφεδρίνη υπάρχει ε, στα φαρμακά και είναι μια ουσία τελείως άχρηστη για τον οργανισμό. Τουλάχιστον στην Τσεχία καταφέραμε να την απαγορεύσουμε. Για τις νέες ψυχοτρόπες λοιπόν ουσίες δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για τα φάρμακα που κυκλοφορούν νόμιμα και μπορούν να γίνουν αντικείμενο καταχρήσεων και ε, και σε μια κουζίνα παράγονται κανονικά τα νέα σύνθετα ναρκωτικά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Σιγητά και φοβούμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε εκείνους που διακινούν αυτά τα προϊόντα τις εγκληματικές αυτές δραστηριότητες, αλλά τουλάχιστον να προειδοποιούμε ένα στον άλλον και να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να τους βάλουμε εμπόδια ή τουλάχιστον να τους δυσκολέψουμε τη ζωή. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I want to the... Ευχαριστώ να καλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο για ε, να μας πει την απόψή της για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ναι, ευχαριστώ από τη μονάδα κατά των στην DG Home η πρόταση αυτή έχει κατόπιν ενός πακέτου δύο προτάσεων που ήδη είχαν υποβληθεί το 2013. Και όπως υπόθηκε επίσης το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να προχωρήσει το προτάσεων αυτών. Η πρόταση που υποβάλαμε τώρα πρόκειται να τροποποιήσει το βασικό κανονισμό του EMCDDA είναι το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που προέκυψε επί Ολλανδικής Προεδρίας και που μας οδήγησε στο να αλλάξουμε την προσέγγισή μας ενσωματώνοντας τις διατάξεις για τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και εξελόγησης κινδύνου στον κανονισμό EMCDDA. Αυτές οι διατάξεις στο παρελθόν <coughs> πρόκειται να συμπεριληφθούν σε μια πρόταση που αφορούσε το άρθρο 113 δηλαδή ως, ε, βάση, ως νομική βάση η αγορά το άρθρο 114 συγγνώμη στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών 2017 λοιπόν αυτό αποτελεί μέρος ενός πακέτου πρόκειται για μια οδηγία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και που επανεξετάζεται από την Προεδρία με βάση το άρθρο 83 της συνθήκης ε, που αφορά το ποινικό δίκαιο θα προλέσει αυτό τη βάση ε, για την όποια δράση αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και να τις ε, θεωρήσουμε ουσιαστικά ναρκωτικά και όπως τα υπόλοιπα ναρκωτικά και να διέπονται από τις διατάξεις. Άκουσα με ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε εδώ ε, στα πλαίσια της μάχης αυτών των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Πρέπει βεβαίως να κινηθούμε γρήγορα. Όπως ε, θα είδατε, στην πρόταση αυτή υπάρχουν πολλά στοιχεία ε, που, έρχεται, που έρχονται να ευθυγραμμίσουν τις διαδικασίες και που μειώνουν τις προθεσμίες ε, και για το EMCDDA αλλά και για, όλους, και για την Κομισιόν, για όλους τους εμπλεκόμενους σε στη διαδικασία αυτή αντιμετώπισης αυτών των νέων ψυχοτραστικών ουσιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα για να κλείσουμε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μπουζόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλίμοβιτ, την κυρία Κονέτσνα, για τις προτάσεις τους ε, αλλά και για το ανοιχτό τους πνεύμα ώστε να βελτιώσουμε από κοινού το κείμενο αυτό αναμένω και από τους λοιπούς σκιώδεις ε, εισηγητές σύντομα θα οργανωθεί μια συνάντηση όπως σας είπα υπάρχει προθεσμία αποβολής τροπολογιών Τετάρτη 19 Οκτωβρίου την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 12 το μεσημέρι μόνο στα αγγλικά οι τροπολογίες παρακαλώ και τον Νοέμβριο θα λάβει χώρα ψηφοφορία η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, είναι καλό το κείμενο. Υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία που είναι απαραίτητα για να ενισχυθεί το σύστημα έγκαιρης και όχι μόνο. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το κείμενο και να μπορέσει να εγκριθεί, να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 10. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, πριν κλείσω το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 12, μόνο στα αγγλικά. 7 ή 8 Νοεμβρίου στην Επιτροπή ΕΝΒΗ θα γίνει η ψηφοφορία, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 17 Νοεμβρίου. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας και από εμάς.